Uh, welcome to the committee meeting. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, έχω δηλαδή μια ιδιαίτερη ανακοίνωση, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, κυρίες και κύριοι, όπως είπα, πρόκειται για μια ειδική ανακοίνωση, πρόκειται για έξτρα συνεδρίαση της Επιτροπής μας μαζί με την Επιτροπή Πολιτισμού, στην βάση του διαδάξεως του άρθρου 55 του κανονισμού. Διότι ε, έχουμε μια κοινή έκθεση. Creating Industries. Δικός μας συζητητής είναι ο κ. Έδερ. Στις 9 Μαΐου, 7 με 9. Το βράδυ φυσικά. Στο Στρασβούργο. Την, την Δευτέρα. Δευτέρα. 7 με 9. Στις 9 Μαΐου. Σημειώστε το σας παρακαλώ, ε, διότι είναι σημαντικό θέμα. Το υπαριθμό 7 τώρα και καλώς ήρθατε όσοι είστε παρούσες και παρόντες για το δεύτερο μέρος της συνεδριάσεώς μας. Όπως είπα, πρόκειται για το θέμα υπαριθμών 7 προς ένα νέο σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας. Με 590 τροπολογίες για την έκθεση αυτή για, που θα θεσπίσει ας πούμε, την πολιτική θέση του Κοινοβουλίου για την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένεται περί τα τέλη του έτους. Άρα είναι, είναι σωστή η χρονική στιγμή για να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο με εισηγητή τον κύριο Λάγκεν, ο οποίος εξετάζει αυτή τη στιγμή τις συμβιβαστικές τροπολογίες που προτίθεται να συζητήσει με τους κοιόδης συζητητές την επόμενη εβδομάδα, εξ όσων γνωρίζω. Αγαπητέ ε, Λάγκεν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να λάβετε το λόγο για να κάνετε κάποιες προκατακτικές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη αναφέρατε τον αριθμό των τροπολογιών. Είχαμε την προθεσμία μέχρι 21 Τρίτου, κατατέθηκε 6 εκατοντάδες περίπου ε, ε, τροπολογιών. Μετά ε, διαβιβάστηκε η συνολική εκδοχή που περιλαμβάνει όλες τις γλώσσες. Αγγλικά υπάρχουν από τις 12 Απριλίου και από την τελευταία εβδομάδα είναι διαθέσιμες πλέον όλες οι μεταφράσεις, ώστε όπως είπατε και εσείς βρισκόμαστε σωστά, ε, βρισκόμαστε χρονικά σωστά. 590 τροπολογίες με πλήθος τροπολογιών μεταξύ αυτών που δεν αφορούν παρά μόνο κάποιες ε, γλωσσικές λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες άρα που ε, επί του ουσιώδους περιεχομένου δεν διαφέρουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορεί κανείς να ενσωματώσει τις τροποποιήσει αυτέ οι οποίε ε, δεν θίγουν την ουσία. Νομίζω το πρόβλημα εδώ δεν είναι μεγάλο. Υπάρχουν όμω, όπω διαπιστώσαμε, και ορισμένα προβλήματα με τις μεταφράσει του γερμανικού κειμένου τη εκθέσεω στα αγγλικά. Θα φέρω ένα παράδειγμα μόνο. Οι διαχειριστές των ε, δικτύων μετάδοσης έχουν μπερδευτεί με αυτούς που διαχειρίζονται τα ε, δίκτυα συνολικά. Και ε, άλλες ε, παρόμοιες διαφορές όρων. Υπενθυμίζω ότι και σε παλαιότερες θητείες καταλήξαμε ορισμένες φορές στην Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενεργείας να μιλάμε παραλλήλως, δηλαδή να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε λόγω των διαφορετικών παραδόσεων ε, σχετικά με το θέμα στις χώρες μας. Τα θέματα ε, επί των οποίων έχουν κατατεθεί αμφιλεγόμενες τροπολογίες είναι αφενός οι μηχανισμοί χωρητικότητας. Εγώ κατέστησα σαφές ότι αυτοί οι μηχανισμοί οδηγούν ή μπορούν να οδηγούν σε στρέβλους του ανταγωνισμού και σε υπεραυξημένες τιμές ενέργειας. Την αντίληψή μου αυτή μοιράζονται πολλοί συναδελφοί μου, ενώ ορισμένες τροπολογίες τάσσονται και υπέρ των ε, capacity mechanisms, όπως οι κυρίες ε, Μπερές, Νίπλερ, Μποναφέ, Μάρτιν. Άρα για το θέμα αυτό θα χρειαστεί να συζητήσουμε να δούμε δηλαδή αν θα έχουν διαμεθοριακό χαρακτήρα, προσωρινό, διαρκή και ούτω καθεξής. Επ' αυτού δημοσίευσε έγγραφο η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είδα εγώ την προσωρινή του εκδοχή χθε και που αναμένεται η οριστική περί τα τέλη του έτους. Πρόκειται για προσωρινή έκδοση για τα capacity mechanisms που θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει μια ορθή συμβαστική γραμμή. Υπάρχουν άλλωστε διάφορες τροπολογίες από τους κυρίους Βένερ, Μπένσεν, Κρέφιν και Σανουάντο. Σύμφωνα με αυτά, οι μηχανισμοί χωρητικότητας θα πρέπει μετά από μια πανευρωπαϊκή ανάλυση της ασφάλειας προμήθειας, αλλά και στο εθνικό επίπεδο, να αποδείχνουν ότι είναι ανάγκη των αγορών. Και ότι είναι ανοιχτή οι μηχανισμοί αυτοί σε όλους τους παρόχους ανεξαρτήτως τεχνολογίας που χρησιμοποιούν. Αλλά εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε για να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Τώρα, η κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά θα πρέπει να επιτρέπονται να ανέρχονται οι τιμές για να μπορούν να δίνουν και μηνύματα οι και οι αγορές. Την αντίληψη αυτή συμμερίζονται πολλοί συνάδελφοι και μάλιστα εξ όλων των πολιτικών ομάδων. Ακόμη και ο Στούρμες Τούρμες στάσεται υπέρ, αλλά και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, κύριος Μπούσεκ, και άλλοι. Ωστόσο, εκφράζουν την ανησυχία οι συναδελφοί μου ότι εκτίθεται σε μη υπολογιζόμενο κίνδυνο οι καταναλωτές και είναι δύσκολο το θέμα το οποίο δεν μπορεί να ε, μετρηθεί πριν από την ε, εκκίνηση πιλωτικών προγραμμάτων. ώστε οι ενεγόμενες αυξήσει τιμών να μην καταλήξουν να επιβαρύνουν τους τελικού καταναλωτέ. Θα πρέπει δηλαδή να μην φτάσουμε στο σημείο να εξετάζουν οι καταναλωτέ κάθε πρωί τι τιμέ του ρεύματο για να αποφασίσουν αν θα ψήσουν καφέ ή αν θα κάνουν τους. Τρίτο θέμα είναι ανανεώσιμε ενέργειε. Στο Κοινοβούλιο έχουμε συμφωνήσει ότι αυτέ θα πρέπει να προωθούνται ε, με διάρκεια και να εντάσσονται στα δίκτυα. Δεν υπάρχουν τροπολογίες που να αμφισβητούν τον στόχο της ένταξης των ε, ανανεώσιμων ενεργειών που έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο της τάξης του 27%, όμως σε διάρκεια χρηματοδοτική ενίσχυση των ανανεώσιμων ενεργειών δεν γίνεται αποδεκτή πλέον από κανένα. Και η αναγκαιότητα της κατά προτεραιότητα διοχέτευσης του ρεύματος από ανανεώσιμες ενέργειες αμφισβητείται πλέον στην στην... Ε, σε ορισμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και στη Γερμανία. Αντί για τι διαρκεί χρηματοδοτήσει, είναι καλύτερα προγράμματα δημοπρασίας βασισμένα στις ανάγκες των αγορών και αυτά να προωθηθούν. Και μόνο εφόσον οι φορεί των ανανεώσιμων ενεργειών αναλαμβάνουν την ευθύνη για το σύνολο του συστήματος, μπορεί τότε να λειτουργήσει η αγορά. Εδώ έχουν υποβληθεί και μια σειρά χρήσιμων τροπολογιών από διάφορους συναδέλφους. Εν προκειμένου, ε, σημαντικές είναι και οι τροπολογίες για την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2014. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Είπαμε, ε, έχετε φτάσει στα 7 λεπτά. Τρία πράγματα μου μένουν ακόμα κύριε Πρόεδρε. Συμφωνείτε να συνεχίσω. Μα πρόκειται για την πρώτη παρουσίαση των τροπολογιών. Πώ είναι δυνατόν στο τέλο τη του. η ευθύνη των κρατών για το μείγμα ενέργειας. Κατά την άποψή μου, όλοι οι φορείς παροχής ενέργειας θα πρέπει να έχουν θέση, την δε ευθύνη θα πρέπει να λαμβάνουν οι χώρες μέλη και να τη διατηρούν για όλα τα είδη ενέργειας. Ακολουθεί ο ρόλος των διαχειριστών των δικτύων διανομής. Εδώ έχουν γίνει τροπολογία την παράγραφο 29, τις οποίες δεν κατανοώ όλες τις τροπολογίες. Τίθεται κυρίως εδώ το θέμα τη διαχειρίσεως των δεδομένων. Τέλος, ο ρόλος της ΕΣΑ. Χαίρομαι που οι περισσότερες και οι περισσότεροι συνάδελφοι συμφωνούν μαζί μου ότι η ΕΣΑ εγκύπτει σε θέματα ασφάλειας προμηθειών και εκεί πρέπει να ενισχυθεί να έχει και την απαραίτητη χρηματοδότηση, να μην αναλάβει όμως μια συνολική εποπτεία της αγοράς ενέργειας. Αντιθέτως, η αγορά να μπορεί να αντιδρά όπως το έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, πολύ ολοκληρωμένη αυτή παρουσίαση. Ο συνάδελφος Ανωνάτος και ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν, σαφώς και πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, ε, καθώς προκύπτει και από τον υψηλό αριθμό των τροπολογιών. Πρώτον, το γενικότερο ε, πλαίσιο της ανακοίνωσης. Το πεδίο εφαρμογή νομίζω ότι εφαρμόζεται καλύτερα με τις ενεργειακές πολιτικές, τις κλιματικές πολιτικές, ε, που είναι αλληλένδετες και θα εξακολουθήσουν να είναι. Οποιοδήποτε ενεργειακό ζήτημα έχει επιπτώσεις και στο κλίμα και το αντίστροφο. Με την ε, πρόταση του εισηγητή, αυτή η πρόταση για την ε, διασύνδεση ενέργειας και κλίματος νομίζω ότι δεν ε, αναδεικνύεται επαρκώς. Και Εάν εξετάσετε το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, νομίζω ότι ε, δεν αξιοποιείται πλήρως. Για παράδειγμα στην πρόταση 22, αλλά και σε άλλα σημεία και από πολλές τροπολογίες, από πολλές πολιτικές ομάδες, ε, ακριβώς ε, θίγεται αυτή η έλλειψη. Δεν αφορά το κόστος της μεταφοράς της ενέργειας. Είναι ένα κέριο ζήτημα, πραγματικό πρόβλημα. και θα πρέπει οι συνομοθέτες να το αντιμετωπίσουν. Το κύριο πρόβλημα, λοιπόν, είναι ότι η ενέργεια και ε, τα κλιματικά ζητήματα είναι αλληλένδετα. Μετά, για τι ανανεώσιμε πηγές ενέργεια. Στι τροπολογίε, έχω προτείνει, όπως και άλλοι συνάδελφοι, μία μη ιδεολογική προσέγγιση ως προς τις ανανεώσιμε. δεν έχουμε βεβαίως και μία προσέγγιση για όλους, one size fits all, ε, στις νέες πηγές ενέργειας. Πρέπει να τα εξετάσουμε βάσει της οριμότητάς τους ε, και της ανταγωνιστικότητάς τους. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην ε, αιωλική ενέργεια ή στα φωτοβολταϊκά. Γιατί να μην εγκαταστήσουμε τέτοιου είδους υποδομές υπερακτίως γιατί η ολική ενέργεια θα εξαρτάται για πολύ καιρό από επιδοτήσεις. Υπάρχει διαφορά μεταξύ χερσαίων και ε, offshore εγκαταστάσεων, υπαρακτήν εγκαταστάσεων. Και όλα αυτά λοιπόν εξαρτώνται και από την ε, δυνατότητα διάθεσή του ε, στην αγορά, τη θέση του σε εμπορία, την ανταγωνιστικότητά τους. Υπάρχουν λοιπόν ε, στοιχεία τα οποία είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια. Και πάλι υπάρχουν ε, διαφορές. Μπορεί κάποιος να εξετάσει το εφιστάμενο ε, πλαίσιο. Δεν μπορούμε να υπερβούμε ή να αντικαταστήσουμε όλους τους εθνικούς μηχανισμούς και εργαλεία. Όμως υπάρχουν κοινά σημεία και εδώ συμφωνώ με τον εισηγητή. Για παράδειγμα, ε, τα εθνικά συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, για, τον, για την ικανότητα παραγωγής είναι κάτι που εξακολουθεί να ισχύει, παρότι κινούμαστε προς μια ευρωπαϊκή αγορά και βλέπουμε ότι οι διασυνοριακές περιφέρειες έχουν ε, πλενασματικό απόθεμα ενέργειας, ενώ άλλοι δεν μπορούν να, τα, να βρουν επαρκή ε, επαρκείς ποσότητες ενέργειας στις δύσκολες περιόδους. Κάτι τελευταίο για την αποθήκευση ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο αναφέρεται σε πολλές ε, τροπολογίες και πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ε, στόχευση ε, στο τι συμβαίνει στην πράξη και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Επομένω, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ. Από την άλλη τώρα, ο κύριος ομιλητής. Ε, ευχαριστώ, λέει ο κύριος Τελίτσκα. Θα μπορούσα να σχολιάσω όλες τις τροπολογίες, ε, αλλά εντάξει, τα ξέρετε αυτά. Μπορώ μόνο να πω ε, δύο λόγια επί της αρχής. Και σε έναν βαθμό βέβαια τα ξέρετε, τα έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Η ουσία είναι ότι η ενεργειακή αγορά αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει τρευλόψεις και νομίζω ότι ο στόχος ε, ενός ανασχεδιασμού της ε, αγοράς ενέργειας είναι κοινός. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν παρέχεται κανένα κίνητρο σε κανέναν να επενδύσει σε οποιαδήποτε ενεργειακή εγκατάσταση. Από πλευράς οικονομικής δηλαδή, από πλευράς τιμών δεν αξίζει τον κόπο. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν ε, χαιρετίζω την έκθεση του κυρίου ε, Λάγκτεν. Ε, Συμμερίζουμε πολλές από τις παρατηρήσεις του. Πολλές από τις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει με τους συνεργάτες μου έχουν ως σκοπό την ακρίβεια, λειτουργούν συμπληρωματικά δηλαδή προς το κείμενο, όμως συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με το γενικότερο πνεύμα, τη φιλοσοφία της πρότασης και νομίζω ότι και το αποτέλεσμα θα αποτελέσει σημαντική συμβολή. Τώρα, θα ακολουθήσω και τη δομή των ε, σχολείων του κ. Λάντεν. Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς ικανότητας, ε, το έχουμε θίξει και εμείς στις ε, τροπολογίες μας. Όντως υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν ιδιαιτερότητες Υπό συγκεκριμένε συνθήκε, ω έσχατη λύση, θα μπορούσαμε ενδεχομένω για ένα μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε τέτοιου μηχανισμού. Θα είμαστε λοιπόν αυστηροί προ αυτό, αλλά θα ακολουθήσουμε τη βασική φιλοσοφία τη έκθεση. Ε, ρύθμιση τιμών. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ε, σημάδια τη αγορά, το οποίο είναι κρίσιμη σημασία. Στο αφορά τη ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, συμφωνώ με όσου λένε ότι οι ΑΠΕ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα επόμενα χρόνια, σίγουρα. Όμω, θα πρέπει ε, να προχωρήσουμε σε άμεση ολοκλήρωσή του. Για το ενεργειακό μείγμα. Και πάλι η ισορροπία που έχει καταφέρει ο εισηγητής είναι σωστή και πρέπει να επικεντρωθούμε σε ζητήματα που θα μας ε, οδηγήσουν πραγματικά σε ένα νέο σχεδιασμό της αγοράς και όχι σε μία διχόνοια. Για τον Acer. Και πάλι θέλουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση για να μην παρεμποδίζουμε ουσιαστικά τον Acer ε, να εκπληρώνει το έργο του. Κλείνοντας, Πρόεδρε, νομίζω ότι το αρχικό προσχέδιο είναι τόσο ποιοτικό που δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν 600 τροπολογίες. Και εδώ παίζουμε με τη φωτιά, γιατί κάποιες τροπολογίες κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αγορά. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Και Όπω είπα, δεν θέλω να επισέλθω σε μεμονωμένες τροπολογίε. Θα συζητήσουμε αυτά με τον εισηγητή και με του υπόλοιπου κοιόδε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στούρμες. Από του πράσινου. Ευχαριστώ πολύ, Τζέρσι. Η αρχική έκθεση αποτελεί καλή βάση. Και εμένα με εξέπληξε το γεγονό ότι έχουμε τόσο πολλέ τροπολογίε. Όμω ε, τα θετικά νέα είναι ότι πολλέ τροπολογίε ε, συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία. Επομένω ε, θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα είναι ευανάγνωστη. Ο κύριος Τελίτσκα έχει δίκιο. Υπάρχει σημαντική εδώ αποτυχία της αγοράς. Ε, η τιμή αυτή τη στιγμή είναι στο 22, 23, 24 σήμερα. Και το ειρωνικό είναι γιατί θεωρούμε ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι 20, 22, 24 λόγω της χαμηλής ε, ικανότητας στην Ευρώπη έχουμε 150 τροπολογίες που ζητούν αύξηση της ικανότητα σε μια αγορά που έχει τεράστια υπερικανότητα, πλεόνασμα ικανότητα. Πρέπει όμω να εξετάσουμε, αν δείτε τι τιμέ, παίζουν καθημερινά, πέφτουν καθημερινά οι τιμέ, γιατί υπάρχει πλεόνασμα ικανότητα. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και την ενδιάμεση έκθεση της Κομισιόν και να είμαστε πιο χαλαροί ως προς αυτό γιατί είμαστε μάλλον υπερβολικοί. Δεύτερον, για την ευελιξία. Η νέα αγορά πρέπει να είναι πιο ευέλικτη. Έχουμε πολλές τροπολογίες ε, για αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι θετικό για τον κλάδο, για τις επιχειρήσεις, τι μικρομεσαίε επιχειρήσεις, τα εμπορικά κτίρια και όχι άμεσα, αλλά μέσω πρόθεσμα και για τα νοικοκυριά. Ασφάλεια εφοδιασμού. Και πάλι δεν πρέπει να είναι ιδεολογική αυτή η συζήτηση. Δεν είναι είτε όλα είναι εθνικά, είτε όλα ευρωπαϊκά. Εγώ πιστεύω στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Και είχαμε και κάποιες καλέ συμβαστικές τροπολογίε σε άλλες εκθέσεις, όπου είπαμε ότι ε, όλους μας συμφέρει η περιφερειακή συνεργασία στο ζήτημα τη άλλη αφοδιασμού, ίσως και εδώ για την αποσύζευξη των ε, TSOs υπάρχει το πρόβλημα ότι το 80% ε, των δικτύων ανήκει μόνο σε 10 επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό σήμερα. Μία πλευρά που εδώ πλέον είναι λογικό το ζήτημα και θα συνεχίσω στα γερμανικά. Πού ε, βρίσκεται η συζήτηση στην Γερμανία επιδοτήσεις της πυρηνικής ενέργειας. Δεν έχετε χρήματα για να καταργήσετε τους σταθμούς αυτούς. Δίνουμε δισεκατομμύρια υπέρ του άνθρακα, ενισχύσει τον άνθρακα. Έχουμε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι δισεκατομμύρια δίνονται στον άνθρακα αντί για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Και μου λες ότι είσαι 110, ε, τον, υπέρ των 110 ευρώ την κιλοβατόρα αντί 70 ε, ευρώ κιλοβατόρα από ανανεώσιμες ενέργειες αυτό είναι απόλυτα ιδεολογικό. Να φανεί σε ρεαλιστή, όπω φαίνεται, σε ρεαλιστή και σε άλλα τμήματα τη εκθέσεω. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Ένστ, ναι, Η κυρία Ένστ. Νομίζω πρέπει να κάτσουμε να κοιτάξουμε με ησυχία τι θέλουμε, με ηρεμία δηλαδή, με, τη νέα, με, το, νέο αυτό σχεδιασμό της αγοράς. Νομίζω ότι όλοι εξ αρχής συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες ενέργειες, έχει καλώς, όμως αυτά πρέπει να τα συνδυάσουμε με τους ε, στόχους για το κλίμα. Αυτό έχει όμως και ε, συνέπειες. Τι γίνεται με τους ε, μηχανισμούς εφεδρείας στις χώρες μέλη. Δεν μπορεί να έχει κανείς το ένα εάν απορρίπτει το άλλο. Γι' αυτό θα καταλήξουμε τελικώς σε αντίφαση. Γι' αυτό νομίζω ότι οι μηχανισμοί εφεδρείας είναι όχι μόνο αναγκαίοι, μάλιστα δεν αρκεί να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντί του, αλλά πρέπει συγκεκριμένα να δούμε τι θα κάνουμε. Οι χώρες μέλη που έχουν την πρόθεση να, το, να τους δημιουργήσουν θα πρέπει να το αφήσουν, διότι πρόκειται για τροχοπέδι για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Αλλά και τα διάφορα μοντέλα που υπάρχουν απανταχού του κόσμου δεν ανταποκρίνονται στις ε, προδιαγραφές για τις ανανεώσιμες ενέργειες και γι' αυτό νομίζω ότι εδώ χρειαζόμαστε μια σαφέστερη διατύπωση. Τώρα, ενεργειακό μείγμα. Ναι, πράγματι αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα, το κατανοούμε κι εμείς, ούτε μπορούμε άλλωστε να το ε, σταματήσουμε, ε, να το οδηγήσουμε σε λήξη. Από την άλλη μεριά δεν θεωρούμε ότι η χρήση όλων των ε, πηγών ενέργειας στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ε, διότι αυτό δεν το έχουμε δει ούτε στην ατομική ενέργεια ούτε στον άνθρακα. Το επόμενο θέμα είναι οι ρυθμιζόμενες τιμές να καταργηθούν και οι διαρκείς επιδοτήσεις επίσης όπως γράφεται εδώ στην εκθεσή σας. Το 2015, επισημαίνω, στη Γερμανία και μόνο στη Γερμανία, 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για επιδοτήσεις πετρελαίου, αερίου και άνθρακος. Το κόστος των ενεργειακών επιδοτήσεων, και αυτό δεν είναι προσοχή έκθεση της αριστεράς, είναι έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όσο υπάρχουν αυτές οι ενισχύσεις, είναι πραγματικά παράλογο να λέμε ότι στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών δεν χρειαζόμαστε ή δεν απαιτούνται επιδοτήσεις. Δεν μιλούμε για διαρκείς επιδοτήσεις, ούτε για επιδοτήσεις κατεσπαρμένες παντού. Ανταυτού πρέπει να επαναξετάσουμε τις κατευθυντήρες γραμμές. Και έχω και μια ερώτηση προς τον εισηγητή για την παράγραφο 23. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε, διότι δεν κατάλαβα πριν καλά, τι γίνεται με τις κυρώσεις. Εμείς λέμε καθαρά όχι στην παράγραφο 25, διότι εκεί επανεμφανίζεται το φάσμα της ατομικής ενέργειας και την προστασία καταναλωτών. Πρέπει να ενισχυθεί. Οι ευφυείς μετρητές έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν μεγάλο αριθμό δεδομένων. Χρειαζόμαστε όμως ξεκάθαρες ρυθμίσεις, διότι με τον βασικό κανονισμό στο συγκεκριμένο αυτό πεδίο δεν προχωρούμε καθόλου. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Ο κύριο Ταμπουράνο που είναι σκιώδη εισηγητής για την ομάδα EFTD. Σας ευχαριστώ να ευχαριστήσω και τον κύριο Λάγκεν για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Να πω κάτι για την αγορά, να πω κάτι για την ενέργεια. Ο σχεδιασμός της ε, ενεργειακής αγοράς είναι κάτι το θεμελιώδες θεωρούμε ότι η Ενεργειακή Ένωση και η ενέργεια μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός συνδετικός κρίκος για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει πριν ακόμα και από το ενίο νόμισμα. Είναι η κινητήριος δύναμη που θα μας επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε, να υλοποιήσουμε πράγματα στην πραγματική οικονομία. Και το κόστος εργασίας και ενέργειας είναι πολύ κοντινέ ενίε. Τώρα, ε, έχουμε διάφορους τρόπους ερμηνείας της έννοιας αυτής. Εμείς θέλουμε μια, ένα ποιοτικό σύστημα που να το εγγυώνται οι δημόσιες αρχές. Και θέλουμε να αποφύγουμε ένα σύστημα στο οποίο κάποιοι ε, κάνουν κάποιες, ε, κάποιες συμφωνίες και κάποιες business σε κάποιους σκοτεινούς διαδρόμους και δεν ενημερώνουν κανέναν. Η ενεργεία είναι η κλίδα για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πραγματική ενεργειακή μετάβαση, αλλά σύμφωνα με τη δική μας ερμηνεία αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τον άνθρακα, από την πυρηνική ενέργεια, από την κεντρικοποίηση. Πρέπει να υλοποιήσουμε από τους, τους στρατηγικούς μας δηλαδή στόχους που περνάνε και από την ενέργεια. Ασφάλεια, ειρήνη, ε, περιβαλλοντική ασφάλεια, οικολογική ασφάλεια, μακαροπρόθεσμα και βιώσιμα. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε μηχανισμούς αγοράς που θα μπορούν να αξιολογούν καλύτερα όλα αυτά, δηλαδή η ανταπόκριση στην ε, ζήτηση και άλλοι μηχανισμοί. Θα πρέπει και όλα αυτά να συμπεριλαμβάνουν έναν υπολογισμό του κόστους του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού, γιατί δάλλως δεν θα ήταν μια πραγματικά ελεύθερη αγορά. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί για τους μηχανισμούς δυναμικού, πρέπει αυτή να είναι μόνο έκτακτου ανάγκης μηχανισμοί και εδώ μπορούν να μας βοηθήσει και το πρόγραμμα καλύτερης διασυνδεσιμότητας μεταξύ των κρατών μελών. Και πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί και η αγορά και το σύστημα θα πρέπει να υπηρετούν τους πολίτες και όχι το αντίστροφο. Ε, γιατί εδώ υπερίσχυσαν κατά την άποψή μας ιδεολογικές τοποθετήσεις που διαχώρισαν την αγορά από τους πολίτες και τους καταναλωτές. Εμείς λοιπόν ζητούμε επιτακτικά και εδώ και καιρό και μαζί με μία αναγνώριση έναν ορισμό. Μία αναγνώριση του συστήματος του, και του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργεί που θα πρέπει να υπηρετεί άπαντες όλους εκείνους που εν πάση περιπτώσει θα επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ενεργειακή μετάβαση. Θα έχουμε χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις και περιβαλλοντικές περιπτώσεις. Αναφέρομαι και στο carbon bubble που το ξέρουμε αρκετοί από εμά. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι εμείς θα μπορούσαμε και να υποστηρίξουμε έναν ισχυρό ρόλο της ε, Κομισιόν ως εγγυητή των σεδικών, δηλαδή στην αρχική της εντολή, στην αφεντική της εντολή ως μεθοδολογικός οδηγός για να οδηγήσει αυτό το σχέδιο να το κατευθύνει. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Σκιώδης, κυρία Κάπελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η έκθεση περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους για τη νέα ε, αγορά ενέργειας και ευχαριστώ τον εισηγητή οι 590 τροπολογίες, έστω και αν ορισμένε, έχουν ως αντικείμενο μόνο ε, γλωσσικές τροποποίησεις, δείχνουν ωστόσο πόσο έντονο είναι το ενδιαφέρον για τον επανεσχεδιασμό της ε, αγοράς ενέργειας. Έχω ορισμένες παρατηρήσεις. Χρειαζόμαστε κοινού κανόνες για όλους όσοι συμμετέχουν στην αγορά ενέργειας. Ε, χρειάζονται ίδιες ρυθμίσεις για όλα τα σχετικά ε, και για τα χρηματιστήρια της ενέργειας και ούτω καθεξής, διότι είναι σημαντικό να εξυπηρετηθεί και το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο της ενέργειας αλλά και άλλα συστήματα. Επίσης, η ασφάλεια των συστημάτων πρέπει να τονιστεί. Οι ανανεώσιμες ενέργειες πρέπει να μπορούν να αναλαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο την ε, διαχείριση του, των συστημάτων. Αυτό σημαίνει οι σημαντικότερες επενδύσεις. Τρίτο, δημοπρασίες για ε, τα ε, δίκτυα. Πρόκειται εδώ για διαφάνεια, για την διασύνδεση και των αγορών. Τέλος, ορισμένα ακόμη σχόλια. Οι όροι του ανταγωνισμού για την χρήση του συστήματος από, συμβατικά, από συμβατικούς παρόχους και με μια συστημική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τους κανόνες. Στην αγορά ενέργειας χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο, σαφές πλαίσιο για όλους τους ε, φορείς που συμμετέχουν στην αγορά. Με καθημερινές δημοπρασίες, το ίδιο σημαντικό είναι να υπάρχουν ξεκάθαρες ρυθμίσεις για τις αποδόσεις των ε, ε, σταθμών παραγωγής ενέργειας ό,τι αφορά την αντιμετώπιση εχμών αυτό πρέπει να γίνεται στη βάση δημοκρασιών σε ηλεκτρονική βάση. Άνοιγμα της αγοράς για τις ανανεώσιμες ενέργειες, για την αντιμετώπιση των εχμών. Και ορισμένα σημαντικά ακόμη σχόλια, τα οποία θα λάβει υπόψη του ο ε, συντάκτης της εισηγήσεως, η ε, προσέγγιση του είναι βασισμένη στην αγορά. Αυτό είναι σημαντικό για να μειωθεί το κόστος και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς αλλά και για την ε, βιομηχανία. Και είναι σημαντικό για να φτάσουμε σε μια πανευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικού ρεύματο. Γνωρίζουμε ότι θα είναι αναγκαίε ε, πολύ υψηλέ επενδύσει για να επιτευχθούν οι στόχοι και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η ασφάλεια προμηθειών. Οι στόχοι των επενδύσεων πρέπει να είναι βασισμένοι στις ανάγκες της αγοράς για να μπορούν να αποδίδουν, πρέπει να επιτραπεί να επιλεγούν ε, καινοτόμες λύσεις, τα μέτρα για, την, για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων πρέπει να είναι επίσης προσαρμοσμένα και τέλος για τους μηχανισμούς δυναμικότητας νομίζω ότι μια λύση επί του παρόντος μπορεί να αποτελέσει η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έχει συμβαστικό χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ κύριος Μπλάνκο Λόπεθ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο αριθμός των τροπολογιών καταδεικνύει το ενδιαφέρον που υπάρχει εδώ και μας προσφέρει μια καινούρια εστίαση που θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας κατά την άποψή μου. Σχετικά με το δυναμικό, σχετικά με την τιμή της ενεργείας και σχετικά με τις επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν. Όπως και σε προηγούμενες ε, τοποθετήσεις, επαναλαμβάνω, ότι το κλειδί βρίσκεται στην ενεργειακή απόδοση, στην καλύτερη αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των ανανεωσίμων πηγών και της ενέργειας που παράγεται από τους ανεξάρτητους πολίτες. Χρειάζεται λοιπόν ανάπτυξη των εφιών δικτύων και υλοποίηση των διασυνδέσεων στην ενωστερική ενέργεια. Με άλλα λόγια, η Ενιακή Ένωση είναι στην ουσία ένα δίκτυο συνδεδεμένης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει ε, προμήθεια σε κατάλληλες συγκρατημένες τιμές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Γκάμπους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκ μέρους της ε, Πιλάρδε Καστίγιο που δεν μπορούσε να είναι παρούσα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τον νέο σχεδιασμό της ε, Ενεακής Ένωσης. Καταρχάς χρειάζεται ένα νέο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και σταδιακή απομάκρυνση από τον άνθρακα, εξασφαλίζοντας όμως την ασφάλεια εφοδιασμού. Δεύτερον, ο στόχος είναι να ανοίξουμε την αγορά κατά τρόπον ώστε οι καταναλωτές να συμμετέχουν ως δυνητική παραγωγή στο πρόγραμμα και να συγκαθορίζουν, να συνδιαμορφώνουν τις τιμές. Και αυτό στηρίζεται σε τέσσερα στοιχεία. Πρώτον, έχουμε ανάγκη για μια αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Πάντοτε σεβόμενοι βεβαίως την ε, κυριαρχία του καθενός για το ενεργειακό μείγμα. Δεύτερον, η αύξηση της ενσωμάτωσης των, των ε, ανανεωσίμων για τις τροπολογίες 16 και 466 αν καλά. Επίσης, χρειάζεται καλύτερη ενσωμάτωση των διασυνδέσεων. Τροπολογία 408, 318 μάλλον. Επίσης χρειάζεται καλύτερη διαχείριση τετάρτων. Ε, τροπολογία 259. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Γκρίφιν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να συνδέσουμε το σχεδιασμό της νεακής αγοράς και τη νέα συμφωνία επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο για τους ενεργειακούς καταναλωτές. Η ενεργειακή αγορά θα πρέπει να συγκρατήσει τις τιμές για τους καταναλωτές και ευχαριστώ τον Φλάβιο για την έμφαση που έβαλε στους ενεργειακά φτωχούς σε αυτή την κατηγορία του πληθυσμού εδώ θα πρέπει να περάσουμε αρμοδιότητα και ισχύ στους καταναλωτές χωρίς να μεταβάλουμε τη συμμετοχή των ανανεωσίμων και ενσωματώνοντας τις καλύτερα στην αγορά. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς ε, ε, αγοράς δυναμικού ή στο ελάχιστο. Αυτές δεν είναι μακροπρόθεσμες λύσεις. Οι μακροπρόθεσμες λύσεις είναι το να περάσουμε την εξουσία στους πολίτες, η ανάπτυξη του δυναμικού αποθήκευσης, όπως είπε και ο Φλάβιο. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε σχετικά με το ρόλο του Acer ότι θα έχει τους επαρκείς πόρους ώστε να αναλάβει τις πρόσθετες αρμοδιότητες που πρόκειται να του δοθούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Oh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Όλιβερ Κόχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την πλευρά μας, με μεγάλη χαρά είδαμε την γενική κατεύθυνση της έκθεσης, γιατί προκύπτει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική σύγκληση σε ζητήματα που στο παρελθόν ε, ήταν αμφιλεγόμενα η σαφή έμφαση στη λειτουργία τη αγορά και στην ε, σημασία τη διατήρηση τη αγορά. διαφαίνεται και είναι πολύ σημαντική. Παρόλες τις πιθανές ε, διχογνωμίες και διαφορε απόψεων σε επιμέρου ζητήματα. Γιατί είναι σημαντικό και ο ρόλο του Κοινοβουλίου εδώ πέρα. Να αποστείλουμε αυτό το μήνυμα ότι δεν πρέπει να επανέλθουμε σε ένα παλαιό ε, μοντέλο ρύθμισης των αγορών ενέργειας. Αυτή είναι η βασική παρατήρηση που θέλαμε να κάνουμε ως προς αυτό το σχέδιο έκθεσης. Για πιο συγκεκριμένα ζητήματα δεν έχουμε δει ακόμα την τελική εκδοχή του κειμένου. Σημεριζόμαστε την άποψη ότι τα ζητήματα που ανέφεραν και οι ομιλητές προηγουμένως είναι αυτά που και εμείς έχουμε εντοπίσει ως ε, ακαθόδη ζητήματα. Από το βαθμό στον οποίο επηρεάζουν οι αγορές ε, ικανότητας μέχρι το βαθμό στον οποίο απαιτείται περαιτέρω περιφερειακή συνεργασία. Και πότε και πού θα βρούμε την ε, κατάλληλη ισορροπία. ανάμεσα στις περιφερειακές αγορές και στους, ε, στην περιφερειακή συνεργασία των TSOs, εν, με παράλληλη όμως διατήρηση των εθνικών αρμοδιοτήτων. και της ε, εθνικής ευθύνης για, την, ε, για τα δίκτυα και το καθεξής. Προς το παρόν, λοιπόν, ε, μπορούμε μόνο να επικροτήσουμε την έκθεση με τη σημερινή της μορφή και βεβαίως στηρίζουμε ε, και την πρωτοβουλία. Thank you much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κάριντ. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ναι, για αυτά που είπε και ο Κλώτ προηγουμένως. Πολλοί από εμά αυτήν την Επιτροπή σίγουρα λειτουργούμε με ιδεολογικό γνώμονα, ανάλογα με την κοσμοθεωρία μα. Άλλοι είναι υπέρμαχοι τη πυρηνική ενέργεια, άλλοι θεωρούν ότι χειρότερο έχει συμβεί στην ανθρωπότητα. Όμω πρέπει να δούμε πώ θα διαμορφώσουμε έναν μηχανισμό τη αγορά που θα αποστέλει τα σωστά μηνύματα και σημάδια για τι κατάλληλε επενδύσει. Γιατί τελικά θέλουμε και καθαρή ατμόσφαιρα και φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, θέλουμε και τι κατάλληλε επενδύσει στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Ο κίνδυνο είναι ότι ω πολιτικοί θεωρούμε ότι μπορούμε με κάποιον τρόπο να νομοθετήσουμε και έτσι να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες επενδύσεις. Όμως αυτό δεν ισχύει. Και αυτό προκύπτει και από το έργο της Επιτροπής. Γιατί τελικά καταφέρνουμε να επανέλθουμε σε παλαιότερες καταστάσεις. Υπάρχουν ακόμα εθνικοί φραγμοί, υπάρχει το θέμα της, ε, των αγορών ικανότητας και υπάρχει αυτή η τεράστια πρόσκληση Ενσωμάτωση ε, των υφιστάμενων ανανεώσιμων. Η ολική, τη υπάρχει, τη ε, δεν υπάρχει, όπως και η ηλιακή ενέργεια. Πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, αυτό είναι το κλειδί. Πρέπει λοιπόν να μην τα εξετάζουμε μόνο από καθαρά ιδεολογική άποψης σε σχέση με την πηγή δηλαδή, αλλά να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε μια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βενερλάγκεν έχει το λόγο για καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ για την συνολικά θετική αξιολόγηση του περιεχομένου της έκθεσης. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους που συμφωνούν με την ε, βασική κατεύθυνση. Ευχαριστώ βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιθυμώ να επανέλθω σε ορισμένα σχόλια ο κύριος Ζανονάτο είπε ότι πρέπει να πράξουμε περισσότερα υπέρ της ε, ενεργειακής πολιτικής και υπέρ της πολιτικής του κλίματος. Ασφαλώς παίζει κυρίαρχο ρόλο και η αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος επιδιώκει πολιτικούς στόχους. Βρισκόμαστε όμως μέσα σε ένα τρίγωνο ανάμεσα στην ασφάλεια προμήθειας, στην φιλικότητα προς το κλίμα και στην οικονομική αποδοτικότητα, δηλαδή τελικώς και στην απασχόληση. Όλα τα θέματα δεν μπορούν να χωρέσουν σε μια έκθεση διότι τελικώς δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο θεωρώ ότι οι ανανεώσιμες ενέργειες δεν επιτρέπεται να αξιολογηθούν ιδεολογικά. Το πιστεύω αυτό, απολύτως. Πρέπει να αξιολογηθούν με κριτήρια αγοράς. Και τότε, εφόσον το πράξουμε αυτό, καταλήγουμε σε απλά ε, συμπεράσματα. Για παράδειγμα, η αιωλική ενέργεια είναι ενεργειακά αποδοτική, η φωτοβολταϊκή όμως όχι. Παρέμβαση ε, ε, τούρμες χωρίς μικρόφωνο. Ε, οι offshore εγκαταστάσεις της Δανίας, για παράδειγμα, είναι ανταγωνιστικές εδώ και καιρό. Υπάρχουν και ειδικότερα θέματα, όπως την ενεργειακή φτώχεια, που πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Είναι όμως άλλες πτυχές, οι οποίες πρέπει να ενταχθούν στο μείγμα ενέργειας ως εθνική ευθύνη. Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους του Άλντε που τοποθετήθηκε μάλλον κριτικά απέναντι στους μηχανισμούς δυναμικότητας. Μα ακόμα και ο κύριος Τούρμες με τον οποίο είχα ήδη μαλώσει για το πρώτο ε, ε, πακέτο για το κλίμα για τα καινούργια οχήματα τα έτη 2007 και 2008 σήμερα έρχεται και με επενή. Κλοντ, κοιτάξτε τι θα σας πω. Είμαι απολύτως κατά των επιδοτήσεων το, για, για τις μεγάλες εγκαταστάσεις στην ε, Μεγάλη Βρετανία, όπου εδώ και μία τριακονταετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιτρέψει ε, μια ελάχιστη τιμή για την απόδοση αυτής της ε, ε εγκαταστάσεως παράγει 4.000 μεγάβατ και που μέσα στα 30 χρόνια έχει φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και πριν να αποχωρήσει ο Αλμούνια, το, το ενέκρινε άλλη μια φορά. Πάλι διακόπτει ο κύριος Τούρμες. Λέει κάτι για τον Επίτροπο Έτιγκερ. Άκου να δεις, ε, η αποφασιστική ε, άποψη ήταν του Επιτρόπου ε, Ανταγωνισμού, του Αλμούνια. Τώρα, η κυρία Έρνστ είπε ότι 49 ε, δισεκατομμύρια δίνονται στη Γερμανία για αέριο, άνθρακα και πετρέλαιο. Αυτά δεν αποδεικνύονται ούτε και από τη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Από αυτά μόνο 2,9 δις είναι άμεσες ενισχύσεις. Κοίταξα τώρα το Δουνουτού στο Google τα υπόλοιπα, τα πέραν αυτού των 2,9 δις είναι εικονικά κόστη που προκύπτουν από άλλα στοιχεία. Αυτά που είπε τώρα ο κύριος Τούρμες για το κόστος της διάθεσης ε, των ε, ε, καταναλωμένων καυσίμων των ατομικών εργοστασίων στην Γερμανία. Έχουμε 20 δις αποθεματικά της βιομηχανίας που διατίθεται για αυτού του είδους την... Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος Μπούζεκ, Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ. Μία τελευταία τροπολογία κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους και θα καταβάλω προσπάθεια κατά το δυνατόν στα πλαίσια των συμβαστικών τροπολογιών να, να ικανοποιήσω το δυνατόν περισσότερους. Όλες και όλους δυσ... θα μπορέσω. Μου είναι αδύνατο να συμβιβάσω κάποιες απόψεις που ε, εν τέλει αποδείχνονται απολύτως αντιφατικές. Ευχαριστούμε ε, όλους τους ε, παρεμβάντες και εισηγητές και εσάς κύριε εισηγητή για τη θαυμάσια αυτή συζήτηση. Έχουμε και το χρονοδιάγραμμά μας. 24 Μαΐου. Περίπου ένα μήνα έχουμε λοιπόν. Δεν είναι δηλαδή και πάρα πολύ ο χρόνο για του συμβιβασμού. Τώρα, το 8. Έκθεση εφαρμογή σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Άλλη σημαντική έκθεση αυτή. Εισέρχεται στη σκηνή ο Μάρκους Πίπερ. Πάλι κάποιες εκατοντάδες τροπολογιών. Ε, αυτή είναι Αυτή είναι η κατάσταση στο Κοινοβούλιο. Δεν έχει μικρόφωνο πρόεδρος. Τώρα έχει μικρόφωνο πρόεδρος. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Πίπερ επεξεργάζεται συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες θα συζητήσει με τους κοιόδης εισηγητάς την επόμενη εβδομάδα. Όπως είπα, αλλά χωρίς μικρόφωνο, παρόλα αυτά θα το επαναλάβω γιατί ήταν σημαντικό, μιλούμε για ενεργειακή απόδοση που είναι πολύ σημαντική για όλες τις πηγές ενέργειας. Τόσο σημαντική και ωστόσο δεν την συζητούμε παρκώς. Κύριε Πίπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες καλές ειδήσει πρώτα. Αφενός έχουμε φτάσει μια εικοσάδα συμβαστικών τροπολογιών και τις 12 από αυτές περίπου τις έχουμε ολοκληρώσει. Ευχαριστώ όλες και όλους που συνεργάστηκαν, αν και καμιά φορά ήταν και πολύ αφιστάμενες οι απόψεις, παρόλα αυτά κάπου μπορέσαμε να ε, τα βρούμε. Μιλήσατε για 330 τροπολογίες για μια έκθεση των τριών σελίδων πάνω από 100 τροπολογίες ανασελίδα. Οι τροπολογίες αυτές μάλιστα προερχόμενες και από κάποιες υπερβολικά δραστήριες πολιτικές ομάδες, ιδίως μία, οι τροπολογίες μιας και μόνης πολιτικής ομάδας φτάνουν τις 40 σελίδες για μια σελίδα της έκθεσής μου. Τα θέτω αυτά υπόψη σας όχι για να κάνω καμιά επίκριση προς Θεού, αλλά διερωτώ με. Είναι δυνατόν να μεταχειρίζεται κανείς έτσι μια έκθεση εφαρμογής εν τέλει. Ποιος ξέρει πόσες συναντήσεις των σκιωδών θα χρειαστούμε μέχρι να τις επεξεργαστούμε όλες αυτές. Τώρα, για την ουσία, άλλη μια καλή είδηση Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε τον στόχο του 20%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε καταρχάς μια πληροφορία που δεν έβαινε προς την κατεύθυνση αρχικώς, αλλά πάντως εάν οι χώρες μέλη συμμορφωθούν, τότε θα επιτύχουμε ίσως μάλιστα και να υπερβούμε τον στόχο του 20% των ανανεώσιμων, κάνοντας έτσι την Ευρώπη πρωτοπόρο στην απόδοση ενέργειας. Φτάνω τώρα στο πρώτο ας πούμε ακαθόδε σημείο όσον αφορά τις τροπολογίες. Δεν είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Αν θέλουμε τώρα περισσότερο μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας υποχρεωτικά ή προτιμάμε την αύξηση της απόδοσης της χρήσης ενέργειας αναμονάδα παραγωγής. Κάτι που δεν κατανοώ από ορισμένες τροπολογίες. Εγώ θέλω να αναφέρω στην έκθεση ότι φεύγουμε από μια οδηγία για την απόδοση ενέργειας και πηγαίνουμε σε μια οδηγία εξοικονόμησης ενέργειας. Ίσως εκεί μπορεί η ε, πολιτική ομάδα να μου εξηγήσει τους στόχους των τροπολογιών της. Τώρα έρχομαι στο θέμα της γνήσιας απόδοσης της ενέργειας. Δεύτερο αγκάθι λοιπόν εδώ είναι το άρθρο 7, υποχρέωση εξοικονόμησης. Πολλοί συνάδελφοι επικρίνουν εδώ ότι οι χώρες μέλη έχουν επωφεληθεί από παράθυρα και από διπλούς υπολογισμούς. Θα χρειαστούν στο μέλλον ξεκάθαροι ορισμοί των δυνατοτήτων που προβλέπει το άθρο 7. Όμως τα εναλλακτικά μέτρα για την ποσοτική υποχρεωτική εξοικονόμηση να παραμείνουν, να εξακολουθήσουν να είναι δεκτά. Εφόσον έχουν γίνει επενδύσεις στην ενέργεια και υπάρχει μια επενέργεια επί της απόδοσης της τάξης των 10-20 ετών, πρόκειται στην πραγματικότητα για μια early action. Δεν αποτελεί παραθυράκι στον νόμο. Είναι μια δυνατότητα που πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται. Τώρα, άρθρο 7. Πώς ορίζουμε αυτά τα παραθυράκια στην νομοθεσία. Εκεί υπάρχουν ποικίλε απόψεις. Έρχομαι στο τρίτο. Αν πόση ώρα μου μένει κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόσεξα το χρονόμετρο. Δύο λεπτά ακόμη. No time at all. Δεν έχετε καθόλου χρόνο. Τότε θα σας πω 7 λοιπόν σχόλια. Καλά λοιπόν, καλά, καλά. Συνεχίζει ο κ. Πίπερ, δυσκολίες αντιμετωπίζουμε και με τις εναλλάξεις δυνατότητες, δηλαδή έχουμε ε, ε, αποδοτική χρήση ενέργειας, eco-design και ούτω καθεξής. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στη βιομηχανία. Αν δηλαδή αλλάξει μια βιομηχανία τον φωτισμό της και βάλει νέας τεχνολογίας, τότε αυτό έχει αποτέλεσμα κάποια εξοικονόμηση ενέργεια. Όμω στι διαπραγματεύσει αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Ενώ θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη αυτή η άμεση ε, επιρροή στο σύστημα εκπομπής καυσαερίων. Τώρα, για τι υποχρεώσει. τέταρτο να Έχω γραπτό πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητούνται από τι χώρε μέλη 200, μπορεί όμως να μπει ένας υψηλότερος πολλαπλασιαστής. Να έχουμε δηλαδή βελτιωμένη συνεργασία και συντονισμό με τις χώρες μέλη, μπορεί τότε και η δράση να είναι πιο συνεκτική. Και αυτή είναι η τελευταία μου σύσταση, δηλαδή περισσότερη συνοχή στην ομοθεσία. Χρειαζόμαστε απόλυτα ξεκάθαρες έννοιες και για τις χώρες μέλη και για τις βιομηχανίες για να επιτύχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση κόστους εν τέλει. Ευχαριστώ να μένω τη συζήτηση. Μύροσλαβ Πόχε. Ο σκιώδης του S&D. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και για την εξαιρετική προφορά. Αγαπητοί συνάδελφοι Σκιώδης, ε, αγαπητοί συνάδελφοι να ευχαριστήσω όλους που υπέβαλαν τις ενδιαφέρουσες τροπολογίες τους. Εγώ θεωρώ ότι η γνωμότητα αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να διαμορφώσουμε μια ισχυρή θέση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. Με την νέα οδηγία που σχεδιάζεται είναι μια μοναδική ευκαιρία να εκφράσουμε σαφέστατα γιατί οι στόχοι που καθορίζει η υφιστάμενη οδηγία κατά πάσα δεν θα επιτευχθούν. Επίσης θα πρέπει να έχουμε προτάσεις όπου το νομοθετικό πλαίσιο θα εφαρμόζεται καλύτερα και θα σχεδιάζεται καλύτερα. Χρειαζόμαστε όμως κάποιες ρεαλιστικές συμβαστικές λύσεις σε κάποια κρίσιμα θέματα. Χρειάζεται να αποστείλουμε ένα μήνυμα στην Κομισιόν για το τι περιμένουμε να συμπεριληφθεί στο σχέδιο της νέας οδηγίας. το παρόν, φοβούμε ότι δεν τα έχουμε καταφέρει με αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή η έκθεση ασχολείται με διάφορα θέματα τα οποία δεν έχουν αγκαστικά επιφέρει την χαμηλή επίδοση που έχουμε στη μέση. Πρέπει να καλύψουμε όλα τα κενά που υφίστανται και ότι δεν θα εκμεταλλευόμαστε την έννοια της ευελιξίας για να μην πληρούμε τις υποχρεώσεις μας. Επίσης δεν υπάρχει μαγική σφαίρα, δεν υπάρχει μαγική λύση στο να επιτύχουμε τους στόχους ενεργειακής απόδοσης. Ε, χρειάζεται ασφάλεια για τους επενδυτές, αλλά ταυτόχρονα όλα τα στήματα στήριξης θα πρέπει να είναι έτοιμα και οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν εμπνευστεί και να εμπιστεύονται τις τεχνολογικές λύσεις που τους προσφέρουμε. Και αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικότητε, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι δυνατότητε των διαφόρων νομοθετικών πλαισίων. Επίση, δεν υπάρχει καμία σύγκρουση με την αύξηση στο ενεργειακό μείγμα των ανανεωσίμων και με το στόχο μα να απομακρυνθούμε από τον άνθρακα. Επίση, για του παραγράφου 15 και 16 να αναφερθώ που αναφέρονται στο πλαίσιο μετά το 2020. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξο και να στοχεύσει σε καλύτερη ενέργεια απόδοση από αυτήν. Προ το παρόν, απέχουμε πολύ από το να έχουμε συμφωνία μεταξύ των σπιωδών επ' αυτού. Αλλά έχει φτάσει η ώρα να βρούμε ρεαλιστικές συμβαστικές λύσεις και υπογραμμίζω κλείνοντα ότι η ενεργειακή απόδοση δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα ανεπιθύμητο άχθος. Αντίθετα, πρέπει να θεωρείται ευκαιρία μοναδική για την βιομηχανία μας και για τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Ντάνκαν δεν είναι παρόν για το ECR. Ποιος θα τον αντικαταστήσει. Δεν βλέπω κανέναν. Άλντε. Ο κ. Πέτρεσεν. Ο Σκιώδης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για μια εξαιρετική δουλειά και τους υπόλοιπους σκιώδεις. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία πράγματι να δώσουμε κάποιες ε, συγκεκριμένες αυτές ενδείξεις για το πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον με τα θέματα ενεργειακής απόδοσης και του συνδεδεμένου φακέλους. Με ικανοποιεί το συνολικό ύφο σχετικά με την υστέρηση υλοποίηση στα κράτη-μέλη και πολύ καλά κάνατε και αναφέρετε το άρθρο 7 πρέπει να συνεχίσουμε να υπογραμμίζουμε το θέμα αυτό ότι δηλαδή θέλουμε επιτυχή και πλήρη υλοποίηση και εφαρμογή των στόχων που έχουμε καθορίσει, θέση πρέπει να εξακολουθήσουμε να είμαστε επικριτικοί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εφαρμογή. και πρέπει να πιέσουμε περαιτέρω. Η αναγνώριση συνεργείας απόδοσης είναι μια πρώτη αρχή. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή κτλ. Επίσης, για τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας που έχουμε προβλέψει εδώ είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και πρέπει να τονίσουμε ότι η οικονομική ανταγωνιστικότητα και η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι σε αντίφαση με, τα, με την ανάληψη μέτρων υπέρ της απόδοσης. Αυτό θα πρέπει επίσης να το υπογραμμίσουμε. Τώρα, έχει γίνει πρόοδος επί μιας σειράς από θέματα. Θα πρέπει ακόμα να επιλύσουμε το δύσκολο ζήτημα της, ευελ... ευελιξίας. Μπορούμε να έχουμε ευελιξία στα μέτρα που επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη, αλλά έχουμε αποκλίνουσες απόψεις για την ευελιξία σε σχέση με τους στόχους. Και δεν θα έπρεπε να είναι εκπληξή ότι εμείς τουλάχιστον είμαστε υπέρ στόχων συνδεμένων με το COP21 με μέτρα ενιακή απόδοση θα πρέπει να τα επιλύσουμε αυτά στη δουλειά που είναι μπροστά μα. Ώστε τελικώ να έχουμε μια έκθεση και μια θέση που να είναι συνεπής και ότι τουλάχιστον συμφωνούμε για το τι εννοούμε με την ευελιξία. Και τι εννοούμε στόχους. Έχουμε όμω πολλέ συναντήσει που τις περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την ερχόμενη εβδομάδα και νομίζω και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι φιλόδοξο και σωστό. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τα σχόλιά σα Από τους πράσινους, σκιώδης συζητητής, ο κύριο Γιάβορ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους σκιώδης ε, για τη συνεργασία τις ε, τελευταίες εβδομάδες. Είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις που περάσαμε, όπως ανέφερε ήδη ο κύριος Πίπερ. Οι απόψεις διήστανται μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων, ωστόσο πιστεύω και εγώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό, τουλάχιστον για τα πιο σημαντικά ζητήματα, για να αποστείλουμε σημαντικό και ισχυρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι κοινό στόχος για όλες τις πολιτικές ομάδες. Μετά υπάρχουν κάποια ουσιώδη στοιχεία της ε, έκθεσης. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Ο κύριος Πίπερ ανέφερε ότι με βάση τις προβλέψεις μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο του 20%, όμως αυτό αποτελεί μόνο δυνατότητα εάν υπάρξει πλήρη εφαρμογή της ε, κείμενη νομοθεσία. Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Και ακολουθούμε μια διαφορετική πορεία που θα μας οδηγήσει πολύ κάτω από το στόχο του 20% με τη σημερινή εφαρμογή. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα, πλήρης εφαρμογή της ε, ισχύουσας νομοθεσίας. Δεύτερον, χρειαζόμαστε και το στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020, βάσει και της Συμφωνίας των Παρισίων και της ε, θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, όπως έχει εκφραστεί σε τρία ψηφίσματα στο παρελθόν, και χρειαζόμαστε και εθνικούς δεσμευτικούς ε, στόχους, γιατί χωρίς αυτό το στοιχείο, στο πλαίσιο μετά το 2020 δεν θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις. Σημαντική είναι και η περαιτέρω βελτίωση της ε, οδηγίας πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση ως προς ε, τα παραθυράκια, την επενδυτική σταθερότητα. Παραθυράκια ιδίως ότι αφορά το σημείο 7.1 πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει πιο λεπτομερείς διατάξεις ε, με ε, ολοκληρωμένους ε, καταλόγους και κατευθύνες γραμμές και δυνατότητες για να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα. Παραμένουν κάποια σημαντικά ακόμα στοιχεία. Νομίζω ότι στην ενεργειακή απόδοση είναι σημαντικά τα σχέδια μικρή κλίμακα, όμω είναι δύσκολο να τα χειριστεί όλα αυτά ακόμα αυτή τη στιγμή. Τα project λοιπόν χαμηλή μικρή κλίμακα θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερου φακέλου, θα πρέπει να αποτελέσει και προτεραιότητα η ενεργική απόδοση ως προς τις κατασκευές και χρειαζόμαστε και την κατάλληλη χρηματοδότηση για να δώσουμε κίνητρα στις επενδύσεις ε, ενεργειακής απόδοσης. Και τελευταίο σχόλιο, νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα για την ε, καταπολέμηση της ενεργειακή ένδυας. Και εδώ χρειαζόμαστε ισχυρή συνεργασία μεταξύ και τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ, σκιώδης, εισηγητής, ο κύριος Βενίτο Ζελουγά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είχαμε σχολιάσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις για την ε, γνωμοδότηση ενεργικής απόδοσης, είναι ένα από τα σημεία κλειδιά για να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σταθερότητα λοιπόν και η δεσμευτικότητα των μέτρων είναι για μας κεντρική σημασία. Και γι' αυτό δεν μας ικανοποιεί το γεγονό ότι και το πρώτο σχέδιο και οι τροπολογίες αφήνουν υπερβολική ευελιξία κατά την άποψή μας για τα κράτη-μέλη προς την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι καλές προθέσεις δεν επαρκούν. Οι στόχοι του άρθρου 7 θα πρέπει να είναι αυστηροί και δεσμευτικοί η παραπομπή στη Συμφωνία του Παρισίου θα πρέπει να είναι πολύ πιο ρητή και συγκεκριμένη και να είναι από τα πρώτα σημεία της έκθεσης κατά την ε, άποψή μας. Αναφέρεται, αλλά όχι με την έμφαση που θα έπρεπε. Και αυτό το σχολιάστηκε και από την Επιτροπή Ένβη. Δεν πρέπει να χάσουμε την οπτική μας από την ε, προσπάθεια αντιστάθμισης και περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και για το αρχικό σχέδιο <clears throat> και στο τωρινό σχέδιο για την προστασία των καταναλωτών και τον έλεγχο της κατανάλωσής τους ή η παραπομπή στην ενεργειακή έμβια σωστά είναι ως σχολεία αλλά δεν είναι επαρκώς τονισμένα όπως έχουμε και εμείς προτείνει σε κάποιες γραπτές τροπολογίες. Επίσης συζητούμε για ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία για να εξωθήσουμε την ενιακή απόδοση. Αυτά ενισχύθηκαν τα στοιχεία αυτά κατά τη φάση διαπραγμάτευσης. Εμείς θεωρούμε ότι η κοινωνική και περιβαλλοντική, δηλαδή κλιματική πτυχή θα πρέπει να είναι πιο σημαντικές διαστάσεις σχετικά. Δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις μας σχετικά με τις ε, δημόσιες επενδύσεις και την συμμετοχή τους στο δημόσιο έλλειμμα που δεν πρέπει να υπάρχει ο συνυπολογισμό δηλαδή αυτό. Δεν θα πρέπει να, έχουμε, να θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πρόσθετο άχθο για τα δημόσια οικονομικά. Ευχαριστώ πολύ. Από το EFDD, ο κύριο Αμπουράνο Να ευχαριστήσω την Αλφό για την προσπάθεια αυτή που κατέβαλε. Διότι εδώ έχουμε διάφορες αποκλίνουσεις, ε, αποκλίνοντα οράματα για το μέλλον και για τον κόσμο. Αναφέρεστε στους στόχους, στα target. Ε, ο στόχος όμως δεν είναι ένας προορισμός, είναι σαν ουτοπία. Είναι κάτι το, το οποίο μας επιτρέπει να προχωρούμε βήμα προς βήμα αλλά να παραμένουμε στο, στο συνεχές παρόν, για να το πούμε έτσι, στο αέναο παρόν. Οι προκλήσεις μας είναι τεράστιες. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του εισηγητή και χρειάζεται ε, συμπόρευση, χρειάζεται κατανόηση. Πρέπει λοιπόν να συμπορευτούμε διότι ακριβώς οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες, τα, δύσκολα είναι, τα προβλήματα μας είναι πολύ δύσκολα και χρειάζεται να συνεργαστούμε. Πρέπει λοιπόν να τοποθετηθούμε σχετικά με το αν αυτό θα πρέπει να είναι ο κινητήριος μοχλός για την αλλαγή ή ένα έρμα, μια τροχοπέδη. Πρέπει να το δούμε ως σταθεροποίηση της κατεύθυνσής μας προ το μέλλον. Χρειαζόμαστε σταθερότητα, ασφάλεια, σταθερότητα για τι επενδύσει. Σε μια εποχή κατά την οποία φαίνεται οι επενδύσει να καταραίουν. Πρέπει να βασιστούμε στην πραγματική οικονομία και οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση επιτρέπουν με εγγύηση των νόμων της θερμοδυναμικής, μάλιστα και όχι δική μας, ε, εγγυημένη κερδοφορία και επιστροφή των επενδύσεων. Ε, χρειάζεται επίσης ε, μια σταθερότητα σε ένα γεωπολιτικό πλαίσιο. Υπάρχουν πόλεμοι γύρω-γύρω μας. Η ενεργεία είναι εξαιρετικά σημαντική με υπό την έννοια ότι όσο λιγότερο εξαρτημένοι είμαστε τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ειρηνικά. Ευχαριστώ. Την ομάδα ΙΕΝΕΦ εκπροσωπεί η κυρία Κάπελ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την καλή έκθεση. Είμαι ε, βεβαία ότι και οι υπόλοιπε τροπολογίες θα ε, μπορέσουν να ε, γίνουν αντικείμενο συμφωνίας τις επόμενες εβδομάδες. Επιτρέψτε μου εν τέλει να τονίσω πέντε σημεία που για μένα είναι σημαντικά. Και στην έκθεση και στις τροπολογίες. Πρώτα, ευκαμψία. 27 από 28 χώρες μέλη αντιμετωπίζουν προσφυγές για παραβίαση της εφαρμογής οδηγίας. Ωστόσο, παρά τις παραβλήψεις αυτές στο επίπεδο των χωρών μελών, έχει επιτευχθεί υψηλός βαθμός εφαρμογής της οδηγίας για την απόδοση ενέργειας. Και αυτό οφείλεται στο ότι και πολίτες και βιομηχανία το επιθυμούν. Παρότι είναι ευθύνη των χωρών, έχει εξασφαλιστεί εν τέλει ασφάλεια των επενδυτών, γιατί είναι μια προσέγγιση βασισμένη στην αγορά. Για το λόγο αυτό και λόγω επίσης των διαφορετικών εθνικών αναγκών, είναι σημαντικό να υπάρξει ένας βαθμός ευκαμψίας και να επιτρέπεται η λήψη και εναλλακτικών μέτρων. Η δημόσια ζήτηση είναι βασικά αυτή που επιβάλλει την βελτίωση απόδοση ενέργεια. Τώρα, υποχρεωτικές υποβολέ εκθέσεων. Για ορισμένες διαμεθοριακώς δραστηριόμενες επιχειρήσεις φτάνουν και παραπάνω από χίλιες εκθέσεις είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν. Αποτελεσματικότητα, τρίτο, δεν σημαίνει απαραίτητα εξοικονόμηση. Αυτό έχει εξηγηθεί και στην έκθεση αλλά και σε ορισμένε τροπολογίε και πρέπει να διατηρηθεί. Σημαντικό είναι ωστόσο να αποφευθούν οι αντιφάσει. Αποτελεσματικότητα τη χρήση τη ενέργεια μέσα στα συστήματα Εφόσον όμως ζητούνται και εξοικονομήσει, πρέπει αυτές να ισχύουν και για τι ανανεώσιμε ενέργειες. Νούμερα και δεδομένα είναι επίσης σημαντικό να συλλέγονται και πέραν των ορίων των χωρών. Με κοινέ προδιαγραφές και για την αξιολόγηση των δεδομένων και για την συλλογή τους. Πρέπει λοιπόν τα δεδομένα να είναι συγκρίσιμα. Αυτό μπορεί να γίνει και εκ των άνω, που βασίζεται όμως σε αόριστες εκτιμήσεις, εκ των κάτω που είναι αρκετά ε, ακριβής αλλά και δαπανηρή και μια υβριδική προσέγγιση που εφαρμόζεται στην πατρίδα μου την Αυστρία και μπορεί να αποτελέσει ένα συμβασμό. Πέμπτον, οι παρεμβάσεις, οι παρεμβολές, διότι αυτά έχουν σχέση και με το εμπόριο των εκπομπών αερίων. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη αυτό. Το λέει και η έκθεση. Και να εξεταστεί ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που οδηγούν στη σημερινή κατάσταση η οποία δεν προσφέρει επαρκή κίνητρα, ε, συγγνώμη, επαρκή κίνητρα για ε, την επένδυση σε ε, βελτίωση της απόδοσης της χρήσης ενέργειας. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, παρά τις 300 τροπολογίες, έχει επιτύχει ευρία, ευρύτατη συνένεση η γνωμοδότηση. Και γίνεται μάλιστα πολύ σημαντική προσπάθεια για την οποία και ευχαριστώ ενσωμάτως των προτάσεων τροπολογίας. Πρέπει κατά την άποψή μας να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στους καταναλωτές και στα συμπληρωματικά κόστη ανατίμησης, ε, στην αναχρηματοδότηση και στις πρακτικές ε, ενεργειακής απόδοσης. Στην παράγραφο 8 λοιπόν για την ε, τροπολογία των 64 υπογραμμίζω ότι τα κόστη που συνδέονται με τις ενεργειακές πολιτικές των κρατών μελών θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν το πλεονέκτημα των τιμών που θα μπορούσε να προέλθει μέσω εξοικονόμηση ενέργειας από τους καταναλωτές. Όσο για την παράγραφο 13 και τον ενεργή ρόλο που θα πρέπει να διαματίζουν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των ε, μέτρων νεαϊκής απόδοσης και για την παράγραφο 10 ότι η ενεργειακή εξοικονόμηση δυσκολεύει την ανάπτυξη των ανανεωσίμων. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λαθασμένο. 78 και 179 που είναι και η δική μου τροπολογία το αναφέρουν αυτό ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Ο κύριος Ζανονάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον κύριο Πίπερ για την εξαιρετική δουλειά. Υπογραμμίζω τα εξής. Αν θέλουμε να δούμε την ε, ενεργειακή απόδοση ως καθαρό καύσιμο, θα πρέπει να αυξήσουμε, να κάνουμε πιο φιλόδοξους τους στόχους μας και θα χρειαστούμε μεγαλύτερη δέσμευση προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό το είχε πει ξεκάθαρα το Κοινοβούλιο και στο τελευταίο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου όπου μιλούσε για δεσμευτικά, δεσμευτικούς στόχους του 40% Επίσης τα ανανεώσιμα θα πρέπει να καταστούν εθνικοί στόχοι. Διότι αλλιώς το λέμε δυνατά, μεγαλόφωνα και μετά δεν γίνεται τίποτα. Για την ενσωμάτωση των εθνικών αγορών στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Κομισιόν μιλάει για περιφερειοποίηση της αγοράς της ενεργειακής απόδοσης και για σταδιακή υπερκέραση των ε, κενών των κρατών μελών και μηχανισμούς ε, ε, απόδοσης δυναμικού. Εδώ θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το λαβύρινθο και την, τη χαοτική αοδό, το χαοτικό αυτό σύστημα, για να πάμε σε μια οργάνωση περιφερειακών και διασυνοριακών κλάστερ. Επίσης η μετάβαση προς ένα πρότυπο ε, οικοσυμβατικού προϊόντος, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα τα οποία τα έχουμε αναφέρει αρκετές φορές αλλά έχουν και κόστος υψηλό κόστος επομένως πέραν από την επιτάχυνση της υλοποίησης της οδηγίας για την απόδειση του 2012 και της ε, οδηγία του 2010 για τα κτίρια θα είναι θεμελιώδε να κοιτάξουμε τα ενεργειακά κονδύλια και ιδιαίτερα το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για να ξεπεράσουμε, να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ Δύσεως και Ανατολής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much, Ευχαριστώ. Η κυρία Κούμπουλα Νάτρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. κρεμούν κάποια ζητήματα από ό,τι κατάλαβα μεταξύ των συντονιστών. Νομίζω ότι πρόκειται για μία έκθεση της πρωτοβουλίας ε, που εξετάζει τα όσο έχουν ήδη επιτευχθεί. Επομένω, πραγματικά σας ε, ενθαρρύνω να σκεφτούμε ε, τι μπορούμε να πούμε στην Επιτροπή και στα κάτι μελη ούτως ώστε να σημειωθεί πρόοδος. Όλοι συμφωνούν μετά για τον στόχο, αλλά το θέμα είναι πώς θα το πετύχουμε τον στόχο. Εκεί θα πρέπει να επεκταθούμε. Στη Φιλανδία, εδώ και 15 χρόνια νομίζω, υπάρχουν εθελοντικά προγράμματα με, το, με τους κλάδους βιομηχανίας που δεσμεύονται από μόνοι τους ε, ως προς τους στόχους ε, περικοπής των εκπομπών και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και νομίζω ότι έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Το ξέρουν και οι επιχειρήσεις, γνωρίζουν το κόστος και στη συνέχεια βέβαια αποτελεί μια εξοικονόμηση για το μέλλον. Είναι λοιπόν ένα στατικό στόχος. Τώρα μετά για ε, τα σπίτια, για τις κατασκευές αλλά και για τα νοικοκυριά. Εγώ έχω ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, και έχουμε υπερψηφίσει αυτό το ζήτημα την περασμένη εβδομάδα με μεγάλη πλειοψηφία, το παρατηρήσατε. Όμως βλέπουμε ότι τα σπίτια μας δεν είναι καλά. Έχουμε ε, τους στίχους, τις κεπές, με διαρροές, με κακή ποιότητας κατασκευή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ενεργειακή απόδοση ωφελεί μόνο τους πλούσιους που έχουν τη δυνατότητα ε, να μετατρέψουν τα σπίτια τους. Πρέπει να έχουμε καινοτόμα μέτρα λοιπόν. Εγώ ασχολήθηκα επί 11 χρόνια στο Εθνικό Κοινοβούλιο με τα ζητήματα και δεν είναι εύκολο όταν έχουμε, όταν έχουμε προγράμματα ε, επιδοτήσεων για τις ε, ανακαινήσεις βλέπουμε ότι οι πιο οικονομικά δύναμοι δεν μπορούν ε, να επωφεληθούν αυτών των προγραμμάτων και μετά πρέπει τέτοια προγράμματα να έχουν στο, και ως στόχο ακόμα και τις ενοικιάσεις ακινήτων για να είναι μόνο οι πλούσιοι που επωφελούνται. Ακούσαμε και από τον Κατάινεν στο Παρίσι για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα έχουμε ακούσει λοιπόν όλα αυτά. Πρόκειται για πιο συγκεκριμένα δηλαδή ζητήματα για μας, για την Επιτροπή Βιομηχανίας, αλλά και πολίτες περιμένουν να, πραγματικά να παρουσιάσουμε έργο. Και για την ευελιξία δεν έχει σχέση με την αποδυνάμωση του κειμένου. Το θέμα είναι να μην ε, απομακρυνθούμε και πολύ από την πραγματική ζωή, το τοπικό επίπεδο, τα σπίτια. Ευχαριστώ πολύ. Άνταμ Γκέρικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εν συντομία, Πρόεδρε. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα έχουμε και πολλές χώρες που θα πετύχουν το στόχο του 20% μέχρι το 2020. Και ο λόγος είναι ότι το λάθος έγινε από την αρχή. Όταν ε, θεωρήσαμε δεδομένο ότι η ενεργειακή απόδοση θα μπορεί να μετρηθεί με φυσικές μεθόδους από τους ίδιους τους καταναλωτές, χρησιμοποιώντας κάποιο είδους εξοπλισμό. Όμως, με τις εξελίξεις στην τεχνολογία βλέπουμε ότι χρειάζονται και κάποιοι άλλοι δείκτες και εγώ προτείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να μας βρουν άλλο τρόπο μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης για όλες τις χώρες. Γιατί αν δούμε τον τρόπο μέτρησης ε, της ενεργικής απόδοσης και στα εργοστάσια και στον μηχανή κτλ, εκεί διαφέρουν τα πράγματα. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Πίπερ. Πρόκειται για έναν ε, περιορισμό ως προς την αξιοποίηση και είναι μάλλον τεχνητό μέτρο. Για παράδειγμα, ανάλογα με το πώς ε, θα μετρήσουμε, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ένα σύστημα είναι εξαιρετικά αποδοτικό, ενώ δεν είναι. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να βρει έναν διαφορετικό τρόπο μέτρησης του βαθμού ενεργειακή απόδοσης. Γιατί αλλιώ βρισκόμαστε σε δύσκολε καταστάσει. Για παράδειγμα, στην Πολωνία βρισκόμαστε στο 17%, αλλά δεν ξέρω αν δεν αλλάξουμε πραγματικά δραστικά τα πράγματα, θα είναι δύσκολο να πετύχουμε το 20%. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο να πάρει τον λόγο από τα μέλη τη Επιτροπή μα. Όχι, από ό,τι βλέπω. Η κυρία Μαρή Ντόνελη, Διευθύντρια από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια, εκπροσωπώντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα μέλη του Κοινοβουλίου για τα επικοινωνικά του σχόλια. Όντω, οι προσπάθειε ε, που έχουν καταβληθεί ε, προ ε, αυτή την έκθεση, όπω είπατε, πρόκειται για μια εξαιρετικά επίκαιρη γνωμοδότηση. Τροφοδοτεί επιπλέον και το προπαρασκευαστικό έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια αναθεωρημένη νομοθετική πρόταση στη συνέχεια τη χρονιά και είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα τα σχόλια των Ευρωβουλευτών δείξατε ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους 2020, όπως ανέφερε και ο εισηγητής, όχι μόνο επειδή και ο κλάδος αλλά και οι πολίτες και οι καταναλωτές στην Ευρώπη το επιθυμούν, επιθυμούν, αλλά και επειδή θεωρούμε ότι σταδιακά η εφαρμογή στα κράτη-μέλη βελτιώνεται. Πράγματι, ξεκινήσαμε με ορισμένε καθυστερήσει και αυτό θα πρέπει να το παρακολουθούμε από κοινού με τα κράτη-μέλη και να υπάρχει συνεργασία μαζί του για να επιταχύνουμε και να αποφεληθούμε το εγχειρήματο. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7, είναι κέρια σημασία ζήτημα, αντικατοπτρίζει 50% των εξοικονομήσεων, συνδέεται στενά και με άλλε νομοθετικέ πράξει, όπω είναι η οδηγία για την αργική απόδοση των κτηρίων, θα αποτελέσουν τμήμα μια ε, δέσμη μέτρων στη συνέχεια. Επομένω, ε, πρέπει αυτό το άρθρο να συνδέεται στενά ε, με την οδηγία λοιπόν για την ειδική απόδοση στα κτίρια, ούτω ώστε και να υπάρχουν οι εξοικονομίε που θέλουμε, αλλά και για να λάβουμε υπόψη και τεχνολογικές εξελίξεις από την υιοθέτηση των δύο νομοθετικών πράξεων και μετά. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο τώρα, μέχρι τώρα οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο ίδιος ο κλάδος ανταποκρίνεται ε, και στις οικονομικές ε, διαστάσεις ε, και το όλο σκεπτικό με θετικό τρόπο και η διάταξη που προβλέπει λογιστικό έλεγχο συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία και πολλές επιχειρήσεις έχουν πει ότι πρόκειται για θετικό στοιχείο. Τώρα, ζητήματα που αφορούν τα κτίρια και στις δύο οδηγίες, όπως είναι τα κίνητρα, δεν είναι εύκολο να επιληθούν η κατάσταση διαφέρει στα κράτη-μέλη, επομένω και οι λύσεις θα πρέπει να είναι διαφορετικές. Όμως, ω προς αυτό, βλέπουμε ότι σιγά-σιγά αρχίζουν να λαμβάνουμε ενδιαφέρουσε προτάσει από τα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη δοκιμάζουν διάφορες λύσεις για το πώς να λύσουν αυτά τα ζητήματα και να βρουν ε, τρόπο επιτάχυνσης ε, του βαθμού ανακαίνησης των ε, κτηρίων που ήδη υπάρχουν, που ξέρετε είναι ένα από τα βασικά προβλήματα. Με τα χαράς λοιπόν βλέπω ότι έχει προσδιοριστεί ο αριθμός των εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται. Το 2000 ήταν υπερβολικό ακόμα και για μας, καλύτερο το 200. Είμαι στη διάθεσή σας, ε, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή άλλη συνδρομή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει και πάλι ο εισηγητή, κύριε Πίπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. και ευχαριστώ όλους όσοι έκαναν ε, πολύ σημαντικά σχόλια. Όντως ε, και οι πολιτικές ομάδες έχουν εξετάσει με μεγάλη προσοχή το ζήτημα. Αυτό το μέσο ε, των εκθέσεων εφαρμογής είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για το Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται μόνο για νομοθετική εργασία λοιπόν, αλλά εξετάζουμε πραγματικά περί τίνος πρόκειται. Τώρα, ορισμένες παρατηρήσεις μιλήσατε για την ενεργειακή ένδυα και πολλοί συνάδελφοι ε, έδειξαν αυτό το ζήτημα. Αν θέλουμε να το καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο, τότε θα πρέπει να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματο. Δεν είναι το υψηλό κόστος τη ενέργειας το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα υπόλοιπα τέλη, χρεώσει ε, ε, με τα οποία επιφορτίζονται οι καταναλωτέ. Και από στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι ουσιαστικά 30% του λογαριασμού της ΔΕΗ, ας πούμε, πάει στο κράτος, 50% στη Γερμανία. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μετά νοικοκυριά που δεν μπορούν καν να πληρώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ και πρέπει από πολιτική σκοπιά να δούμε τι πρέπει να αλλάξει. Η ενεργειακή ένδια λοιπόν το έφυξε και η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να λάβει κεντρική σημασία στην έκθεση. Δεύτερο σχόλιο υποχρεωτική εξοικονόμηση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν ε, θα εμποδίζει άλλα στοιχεία. Όλοι θέλουμε να μεταπηδήσουμε, για παράδειγμα, στα, στις ηλεκτρικές μπαταρίες, στα αυτοκίνητα, με υποχρεωτικό τρόπο. Όμως, Και αυτό θα έχει μεγάλο κόστος. Θα απαιτείται μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Και δεν ξέρουμε αν έχουμε την αντίστοιχη ικανότητα. Δεν γίνεται λοιπόν και να λέμε ότι θέλουμε να μετοποιησουμε στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και να κάνουμε εξοικονόμηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτείται λοιπόν μια συνέπεια εδώ πέρα. Πρέπει λοιπόν να συμβαδίζουν τα όσα λέμε και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Επιτροπή να το εξετάσει περαιτέρω. Κάτι τελευταίο, Πρόεδρε, το αναφέρατε και εσείς στην αρχή. Η ενεργειακή απόδοση ως ε, καλύτερη αρχική πηγή ενέργειας. Πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας, νομίζω. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ε, εντάξει, σίγουρα. Δεν υπάρχει κάτι το ιδανικό παρότι τίνουμε να μην το πιστεύουμε. Η ενέργεια βασίζεται στους πόρους, επομένως πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο ακολουθούμε τη σωστή προσέγγιση και κατά πόσο ε, στέλνουμε το κατάλληλο μήνυμα προς την ενεργειακή απόδοση. Πρέπει λοιπόν ε, να λειτουργήσουμε έγκαιρα, ρεαλιστικά, και με γνώμονα τα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ζηγητή για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Συμφώνησαν σχεδόν όλοι οι σκιώδεις. Και τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Ψηφίζεται στην Ήτρε στις 24 Μαΐου Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σα για τι συμβαστικέ τροπολογίε. Στην Ολομέλεια θα ψηφιστεί στις τον Ιούλιο του 2016. Σα ευχαριστώ όλου. Σημείο 9. Έκθεση προόδου για τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Η συνάδελφος Παλώμα Λόπεθ Βερεμέχο από την ΚΟΕ έχει το λόγο ως εισηγήτρια. 345 τροπολογίες βλέπω. Η προθεσμία αποβολής τροπολογιών εξέπνευσε πριν από μερικές ημέρες. Και τώρα περιμένουμε τη μετάφραση. Αυτή η έκθεση διάσπρωτοβουλίας θα μας ενημερώσει για τα όσα έχουν ήδη γίνει, αλλά και τα όσα θα γίνουν στο μέλλον, ε, ε, εν ώψη του στόχου του 2030. Πλέον δηλαδή σκεφτόμαστε τι θα γίνει με τον ορίζοντα 2030. Η συγγήτρια επεξεργάζεται συμβαστικέ τροπολογίε και θα συζητάει όλα αυτά με τους κοιόδες. Συνεχίζεται η συζήτηση από ό,τι κατάλαβα. Κυρία Λόπεθ Μπερμέχο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, 345 τροπολογίες και προσπαθούμε να βρούμε μια συμβαστική λύση και να το κάνουμε αυτό συλλογικά. Και από αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας για μια ακόμα φορά την προσπάθεια όλων των ομάδων που μας απέστειλαν σε τόσο στενό χρονοδιάγραμμα τις τροπολογίες τους για να μπορέσουμε να επιτύχουμε συμβαστικές λύσεις. Γνωρίζουμε τη στενότητα του χρονοδιαγράμματος, γνωρίζουμε τη φιλοδοξία ώστε να έχουμε ολοκληρώσει πριν το καλοκαίρι με την έκθεση αυτή. Τώρα, υπάρχει μια συνένεση σε πολύ ουσιαστικά ζητήματα, μια συνένεση που ελπίζω να μπορέσει να μεταφραστεί σε σημαντική στήριξη και πλειοψηφική στήριξη. Και αυτό δεν το λέμε, μάλλον. Πρέπει να κοιτούμε και το παρελθόν, όχι για να κοιτούμε το παρελθόν, αλλά για να ετοιμάζομαστε για το μέλλον για το ποια θα πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή πολιτική ανανεωσίμων. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η έκθεση να εντοπίζει, να καθορίζει τις χώρες που έχουν μείνει πίσω αν θέλετε. Αυτό το συζητούσαμε ήδη από την προηγούμενη συνεδρίαση. Θα πρέπει να απαριθμούμε και να καθορίζουμε και εκείνες χώρες που είναι παραδείγματα, υποδείγματα προόδου έχουμε διαφορετικά εθνικά πρότυπα και αυτό είναι σε κάποιο βαθμό φυσιολογικό. Και οι πολιτικές ε, παραγωγής είναι κρατικές και επομένως εθνικές. Πρέπει να δούμε όμως ποια μοντέλα, ποια πρότυπα λειτουργήσαν στο παρελθόν και γι' αυτό μιλούμε για το παρελθόν και ποια όχι. Χρειαζόμαστε ένα σταθερό ρυθμιστικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι θέμα κλειδί για του επενδυτέ. Δεν το εξασφάλισαν όλε οι χώρε αυτό. Χρειαζόμαστε διευκρίνηση των αρμοδιοτήτων. Να μην υπάρχει ασάφεια εκεί. Και θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον τα συστήματα, αν θέλετε, ανακατανομής των ανανεωσίμων πηγών θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες χώρες που υπήρξαν υποδειγματικές μέχρι στιγμής για την παραγωγή και τη διάχυση της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει τους, τις δομές της, της επιτήρησης και παρακολούθησης και να ενισχύσει τη συνεργασία της με κράτη-μέλη. Μιλούμε για συνεργασία με τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να ενισχύεται και με μια ευρύτατη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων, των κοινωνικών φορέων, των τοπικών φορέων, των οργανώσεων καταναλωτών και μη καπαόμικρων. Ο ρόλος όλων αυτών των συμμετεχόντων φορέων θα είναι θεμελιώδης, γιατί έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις οικονομικές, κοινωνικές, εργασιακές, περιβαλλοντικές που μας επιβάλλουν μία ενεργειακή μετάβαση δίχως την οποία δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους του Παρισιού τους οποίους πρέπει να θεωρούμε δεσμευτικούς και με κανέναν άλλο τρόπο. Επομένως, έχουμε ε, ευχαριστήσει ήδη την Επιτροπή Περιβάλλοντος για τη δική της συνεισφορά, αλλά εδώ μιλούμε για μια μετάβαση με τρόπους παραγωγής πιο αποκεντρωμένους, πιο δημοκρατικούς, πιο συμμετοχικούς, απέναντι στις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και, και μόνον έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχουμε απέναντί μας ώστε να έχουμε μια πραγματική συμμετοχή των πολιτών της κοινωνίας και στην παραγωγή και στην κατανάλωση και στην αποθήκευση της ενέργειας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μπέντσεν που εκπροσωπεί το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον ε, εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία, την εισηγητρία, παρότι δεν συμφωνούμε σε κάποια πολιτικά ζητήματα. Ωστόσο βέβαια όλοι κατανοούν την αξία μιας ευρύτερης πολιτικής συνεννόησης εδώ. Εν μελλοντικών εκθέσεων. Για την Ενεργειακή Ένωση επίσης θα ήταν πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε από αυτού γρήγορα, ταχύτατα. Και εν ώψη της ε, εκθέσεως της Επιτροπής του Φθινοπόρου. Εμείς εστιαστήκαμε στα πιο σημαντικά από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικότητα κόστου ωφέλου. χρειαζόμαστε στοιχεία που θα οθούνται από την αγορά, που θα στηρίζονται στην αγορά. Και θεωρούμε ότι η πρόοδος δεν είναι αρκετά ικανοποιητική αυτή που έχει γίνει για τις ανανεώσιμες. Θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια, χωρίς όμως να θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν, να δείξουμε κάποιον με το δάχτυλο. Αλλά εφόσον επιθυμούμε να ενσωματώσουμε ένα καλύτερο μείγμα ένα αυτό εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη, αλλά κυρίως θα πρέπει να δώσουμε στον καταναλωτή πρόσβαση σε ενδιαφέρον ε, ενεργειακό μείγμα, το οποίο θα είναι και ελκυστικό και ενδιαφέρον υπό την οικονομική έννοια. Και ε, υπογραμμίζουμε το θέμα της αποκέντρωσης το οποίο όμως υπό κάποιες έννοιες δεν είναι απόλυτα θετικό. Και εδώ αποτυπώνει τις ε, πολιτικές κατευθύνσεις της συζυγήτριας. Η αποκέντρωση μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική, όταν όμως έχει μια κατεύθυνση και όταν δικαιολογείται και υποστηρίζεται από επιχειρήματα. Συνδέουμε μια συγκρατημένη λογική τιμή στην αγορά και μία, και μία παραγωγή ιδιωτική, θεωρώντας ότι η αποκέντρωση θα έχει μικρότερο οικονομικό κόστος. Ε, συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να συγκρατηθούν, ότι πρέπει να μειώσουμε το επίπεδο της εξάρτησης της ενεργειακής. Αλλά θα πρέπει και οι ανανεώσιμες τιμές να αντιστοιχούν σε ένα πραγματικό, αληθινό οικονομικό κόστος. Και πρέπει να δούμε και το θέμα της βιωσιμότητας ε, των ε, ανοσίμων πηγών. Εν πάση περιπτώσει είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια για να αναπτύξουμε ευρύτερους, ε, ευρύτερους συμβασμούς και συνεννόηση. S&D λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μόλναρ. Köszönjük a munkáját jelentéstevő asszonynak láthatóan az esetek többségében. Ευχαριστώ, Να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια που έλαβε υπόψη μας ε, τι ε, αρκετέ τροπολογίε. είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε συμβαστικέ που θα βρίσκουν σύμφωνες τις πολιτικές ομάδες. Θα επικεντρωθώ τώρα ε, σε εκείνες επί των οποίων δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα. Το δεσμευτικό των στόχων καταρχάς για την περίοδο μετά το 2020 για την ποσόστοση της, ε, των ανανεωσίμων. Όλες οι εκθέσεις και η εμπειρία της Κομισιόν μας δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο στις ανανεώσιμες στην Ευρώπη διότι όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε εθνικό επίπεδο καθορίσαμε δεσμευτικούς στόχους, τους οποίους θα πρέπει να τηρούν τα κρατημέλη. Έτσι εξασφαλίζεται η προβλεψιμότητα, εξασφανίζεται η ανάπτυξη οικονομική. Γνωρίζουμε ότι ακόμα αυτό είναι αντικείμενο ε, συζήτησης εντός του ΕΛΚ αλλά χωρίς δεσμευτικούς στόχους δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε στόχους για το μέλλον έτσι όπως το επιτύχαμε μερικώς και για το παρελθόν. Τώρα υπήρξαν κράτη-μέλη που είχαν, ε, αν θέλετε, επιδόσεις λιγότερο εντυπωσιακέ από άλλων κρατών μελών. Η Κομισιόν θα πρέπει λοιπόν να μας πει ποιες είναι αυτές οι χώρες και πώ θα μπορούσαν να καλύψουν το χάσμα που τις χωρίζει από τις πιο προχωρημένες. Και βεβαίω το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τα εύσημα και στις χώρες που επέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα. Διότι εκτό από τις δεσμευτικέ ε, υποχρεώσεις ανέλαβαν και κάποιες ε, συμπληρωματικέ πρωτοβουλίες προφανώ για να το κάνουν. Τώρα για το νομοθετικό πλώσιο για τις ανανεώσιμες και από πλευράς μας υποβλήθησαν Πολλέ ε, ε διότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, χώρες που έχουν ένα επίπεδο φορολόγηση τέτοιο που αποφέρει ε, οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς. Εμείς είμαστε σαφώς κατά τέτοιων στρεβλωτικών επιβαρύνσεων. Ένα τέταρτο ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε είναι η ενεργειακή ένδυα. Εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι εκ του γεγονότος ότι η συγκήτρια έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα αυτό. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει ένα επίπεδο ευζοίας που το ζηλεύει ολόκληρος ο κόσμος και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχουν χιλιάδες χιλιάδων άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποβαίνουν από ενεργειακή φτώχεια. Που θα πρέπει να επιλέξουν δηλαδή αν θα θερμάνουν το δωμάτιό τους ή όχι. Είναι σημεία που αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε μία νύχτα. Αλλά πρέπει να δούμε την καλύτερη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων με τα κρατημέλη και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα να εξαφανίσουμε το φαινόμενο της ενεργειακής ένδυας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι εκκρεμούν ακόμα συζητήσει, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι η συγκέντρια θα μπορέσει να επιτύχει μια πολιτική συμφωνία για να έχουμε ευρύτατη πλειοψηφία υπέρ τη εκθέσεω αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Βαμπόσφατ από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η τρίτη φορά που εξετάζεται αυτή η έκθεση στην Επιτροπή μας. Όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου είχαν ενταξύ τη δυνατότητα να αναφέρουν τις απόψεις τους ε, ως προς ε, το προσχέδιο που μας ε, παρουσίασε η συγγήτρια. Εμείς θέλουμε πραγματικά με τις τροπολογίες μας να καταστήσουμε αυτή την έκθεση μια έκθεση πραγματικά της Ήτρε. Η εισηγήτρια επικεντρώνεται κυρίως στην κοινωνική διάσταση ε, της ενέργειας, όμως ε, και στο Στρασβούργο ψηφίσαμε την ε, σχετική έκθεση. Πρέπει λοιπόν τώρα να επικεντρωθούμε στην ουσία του ζητήματος. Γι' αυτό θα πρέπει να τηρήσουμε και την αρχή της επικουρικότητας και να θέσουμε τις βάσεις για το νομοθετικό έργο που μας περιμένει στη συνέχεια της χρονιάς. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους να αποφύγουν το φαινόμενο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, δηλαδή τη υπερφόρτωση ε, τη έκθεση με επιμέρου στοιχεία. Τώρα, ορισμένε παρατηρήσει. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο εφικτό των ε, στόχων που θέτουμε. Χαιρόμαστε που η συγκήτρια έχει λάβει υπόψη αυτή την έννοια και στο πρώτο προσχέδιο κατόπιν ε, των τροπολογιών. Δεύτερον, οτιδήποτε έχει σχέση με τη φορολόγηση θεωρούμε ότι είναι μάλλον είναι εθνική αρμοδιότητα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επεκταθούμε ε, αένα σε αυτό το ζήτημα. Τρίτον, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω ότι πετυχαίνουμε αυτό το στόχο μας, επομένω να ε, επικεντρωθούμε κυρίως στην θέρμανση και ψήξη και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τους κλάδους όπου τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, ας σταθούμε περισσότερο σε αυτούς ε, που υπολείπονται. Τέταρτο σημείο, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ε, να ενθαρρύνουμε στην ενέργεια στο πλαίσιο της ενιαίας λειτουργίας αγοράς. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να πείσουμε ε, ότι είναι κάτι το ωφέλιμο και απαραίτητο. Χαίρομαι που επιτέλους ε, μπαίνουμε στην ουσία και μπορούμε να ε, επεξεργαστούμε καλές συμβαστικές τροπολογίες βλέπω σε συνεργασία με την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους κοιόδης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βαν Βόσχατ για τις παρατηρήσεις σας. Εξ ονόματος της Άλντε, ο κύριος Γερμπράντη, σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για το έργο της μέχρι τώρα και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε στις επόμενες εβδομάδες να βρούμε και συμβαστικές λύσεις. Ξεκινώντα, θα ήθελα να πω ότι αν γέννη τείνουμε να είμαστε αρκετά επικριτικοί ω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Όμω, να ομολογήσουμε ότι είναι ένα εξαιρετικά επιτυχή ε, τομέα πολιτική βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας ως προς τις ΑΠΕ μέχρι το 2020, τουλάχιστον ε, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στι μεταφορές υπάρχουν μεγαλύτερε δυσκολίες για να πετύχουμε τον στόχο του 10%, αλλά εντάξει, τουλάχιστον μπορούμε να, να είμαστε αισιόδοξοι ότι βρισκόμαστε στη σωστή τροχιά. Και αυτό είναι σημαντικό σημείο κίνηση. Δεύτερον, πρόκειται για μια έκθεση προόδου και αφορά την κατάσταση που επικρατεί στα κρατημέλη. Είναι λοιπόν ε, παράξενο να πει κανεί ότι δεν πρέπει να κατανομάζονται τα κρατημέλη, γιατί ακριβώ θέλουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κρατημέλη. μελη Επομένω, εννοείται ότι πρέπει να αναφέρουμε και τα κρατημέλη που ε, πηγαίνουν καλά και τις, υπόλοιπε τις υπόλοιπες ε, χώρες που δεν πηγαίνουν τόσο καλά. Όπως η δική μου, οι κάτω χώρες που βρίσκεται κάτω-κάτω στον κατάλογο ε, σε ό,τι αφορά τις χώρες ε, που αξιοποιούν τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μία γενικότερη παρατήρηση. Πάνω από 300 τροπολογίες νομίζω έχουν υποβληθεί. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε ένα σημείο εστίασης, γιατί μια τέτοια εστροπολογιες νομιζω εχουν υποβληθει έχει πολιτική επιρροή μόνο αν έχει συγκεκριμένη στόχευση και θέτει προτεραιότητες. Ας μην επεκταθούμε σε πάρα πολλά ζητήματα, ας επικεντρωθούμε στα πλέον σημαντικά. Ας αναφέρω ορισμένα. Consumers, prosumers. Είναι σημαντικό να καθορίσουμε τον ε, ρόλο τους ε, και τους, για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς καταναλωτές λοιπόν. Αλλά να είμαστε συνεπείς και με την άλλη έκθεση ε, για τον ρόλο των καταναλωτών στην ενεργειακή αγορά. Ας μην επαναλαμβάνουν λοιπόν τις προσπαθίες μας. Για τον τομέα των μεταφορών έχει ήδη αναφερθεί ότι το 5,7% που βρισκόμαστε σήμερα δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικό. Το ανέφερα προηγουμένω. Αλλά α μην είμαστε και υπερβολικά επικριτικοί σε ό,τι αφορά το βιοκαύσιμα. Και νομίζω ότι η συγγήτρια ήδη κάνει λόγο για αποτυχία στο σχέδιο έκθεση. Νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολικό. Τα όσα κάνουμε αυτή τη στιγμή, ιδίω για τα καύσιμα δεύτερη γενιά είναι πολύ σημαντικά. Και για να είμαι ειλικρινή, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει η λύση στον τομέα των μεταφορών αν είμαστε προβολικά επικριτικοί ως προς τα βιοκαύσιμα. Σίγουρα θα πρέπει να θέσουμε κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα, όμως ας μην αποκαλέσουμε αυτή τη στιγμή το σύνολο της πολιτικής μια αποτυχία. Μετά, για την ενεργειακή ένδυα, εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Για μένα συνδέεται περισσότερο με το προηγούμενο ζήτημα που εξετάσαμε, την ενεργειακή απόδοση και όχι τόσο με τις ανανεώσιμες. Και στο παρελθόν έχουμε δει ότι ε, τα καθεστώτα ενισχύσεων για την ενεργική χρήση αξιοποιούνται μεν από τους ε, φτωχούς, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό αξιοποιούνται από τους ε, πλουσιότερους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τέτοιου είδους ε, συστήματα ενισχύσεων. Πρέπει, πιστεύω, καλύτερα να επικεντρωθούμε στην ενεργειακή απόδοση και μετά στο μέλλον καθώς θα αυξάνεται το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πέφτουν και οι τιμές. Εκεί θα είναι το όφελος, πιστεύω. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση προόδου της επίσης καλεί και τα κράτη-μέλη να αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τους το μηχανισμό συνεργασίας. Νομίζω ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη επιμένουν σε έναν ε, εθνικιστικό τρόπο προσέγγισης. Πρέπει να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία και αυτό θα μας ε, βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό και να πετύχουμε τους ε, στόχους μας για το 2020, αλλά και μετά για το 2030. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε, ο κύριος Διάβολο, σκιώδης ηγητή των Πράσινων. Στα αγγλικά σα ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους Σκιώδη για την συνεργασία. Επί του παρόντος, στην εξέλιξη του Έχουμε συζητήσει γενικά θέματα και όχι ειδικέ τροπολογίες. Γι' αυτό και θέλω να έρθω σε ορισμένα γενικά θέματα που έθεσε ο εισηγητής σε προηγούμενες συναντήσεις μας. Πρώτα, θα αναφέρουμε συγκεκριμένες χώρες σε ό,τι αφορά την αποδοσή τους ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να με τις χώρες εκείνες που καθυστερούν, διότι στόχος της εκθέσεως πρόοδου είναι ακριβώς να τονίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά και να δείξουμε και πού είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι πολιτικές, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά μέρη της εκθέσεως, για να αναδείξουμε πού πρέπει να καταβληθούν περισσότερες και εντονότερες προσπάθειες. Δεύτερο, εθνικοί στόχοι. Χρειαζόμαστε εθνικούς στόχους για το 2030 ή όχι. Εγώ πιστεύω απολύτως ότι χρειαζόμαστε. Οι εμπειρίες της οδηγίας για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, η αποδοτική χρήση της ενέργειας και για τις ανανόσιμες ενέργειες δείχνουν σαφώς ότι τα όσα πετύχαμε ως τώρα βασίζονται ιδίως στους εθνικούς στόχους για τους οποίους είναι υπεύθυνε ή χώρε μέλη. Τρίτο θέμα, αναδρομικά μέτρα, ιδίως για τι επενδύσει σε ανανεώσιμες ενέργειε. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένα ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο να είναι προβλέψιμο. Και είναι αναπόφευκτο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο Τέταρτο θέμα, ο ορισμός των παραγωγών καταναλωτών. Πιστεύω ότι αυτοί βρίσκονται στην καρδιά των μελλοντικών συστημάτων ενέργειας στην Ευρώπη. Ιδίω για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεπώς νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε μια κοινή έννοια των παραγωγών καταναλωτών και να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο να στηρίζει τους παραγωγούς καταναλωτές ώστε να γίνουν πιο ενεργά συμμέτοχοι στην αγορά ενέργειας. Τέλος, να μιλήσουμε για συγκεκριμένους τομείς. Μιλούμε για ανανεώσιμες ε, ενέργειες, μιλούμε για μεγάλες εγκαταστάσεις, αλλά από την άλλη μεριά ε, θέρμανση και ψήξη, νοικοκυριά, εγκαταστάσεις αποθήκευσης κλπ. Είναι επίση πολύ σημαντικά τμήματα του θέματος. Άρα πρέπει να μας απασχολήσουν και αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Ταμπουράνο, που θα είναι συγγητής την επόμενη φορά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω ότι ήταν χαρά που συνεργαστήκαμε με την Παλώμα είχαμε έναν σαφή διάλογο και μπορέσαμε να συζητήσουμε ιδιαίτερα επί των κοινών μας, ε, κοινών μας σημείων. Αναφέρθηκαν και άλλοι συναδελφοί στην ενεργειακή φτώχεια και δεν θα ήθελα να επαναλάβω. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια άλλα στοιχεία. Καταρχά, για μας είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να συζητούμε σοβαρά για, τον, για την έννοια των prosumers, δηλαδή των παραγωγών καταναλωτών. Χωρίς ένα κοινό ορισμό, ιδιαίτερα εν ώψη των μελλοντικών νομοθετικών φακέλων, δεν μπορούμε να αναφερόμαστε, να αναφέρουμε τον όρο αυτό έτσι, prosumers, χωρίς να τον ορίζουμε. Και τι μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε ε, την συμμετοχή τους στην αγορά ενέργειας πώς θα μπορέσουμε να καταγράψουμε τα όποια κενά των καταμετρήσεών μας, της παρακολούθησής μας. Στην νέα οδηγία θα πρέπει να υπάρχει ένα κεφάλαιο που να αναφέρεται εις τους παραγωγούς ε, καταναλωτές. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους από τους πράσινους ε, για να έχουμε έναν ορισμό και για τον παραγωγό καταναλωτή τον επαγγελματία. Σε κάποια κράτη-μέλη, στην Ιταλία, στην Ισπανία και φαντάζομαι και σε άλλες χώρες, έχουμε μια τάση χρησιμοποίησης των, από των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες, ώστε να παρεμποδίσουν την εξέλιξή τους και την ανάπτυξή τους. Αυτό εμποδίζει και ζημιώνει την ε, ανταγωνιστικότητά μας και τις ε, επενδύσεις. Εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα πρέπει να το ξαναεξετάσουμε και να το βελτιώσουμε. Όχι να το αποσύρουμε και να το καταργήσουμε. Και οι τράπεζες λειτουργούν κακά μερικέ φορές αλλά εξακολουθούμε να τις βοηθούμε και να τους δίνουμε τα χρήματά μας. Εμείς λοιπόν για τη νέα οδηγία για τα ανανεώσιμα ζητούμε ένα στόχο 45% για το 2030 το οποίο θα πρέπει να αναλύεται σε δεσμευτικούς στόχους εθνικούς. Στόχους που δεν πρέπει να τους βλέπουμε ως ε, βαθμολογία, αλλά ως βήματα απαραίτητα για να φτάσουμε σε μια οικονομία που θα έχει ενσωματώσει τα ανανεώσιμα, που θα έχει αλλάξει σελίδα, θα έχει περάσει το μέλλον δηλαδή. Χρειαζόμαστε λοιπόν φιλόδοξους στόχους που μας δίνουν μια ελπίδα για το μέλλον χωρίς να μένουμε σε ένα φαιό παρόν που δεν κινούμαστε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Τζανονάτο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η συγγήτρια σωστά υπογραμμίζει ότι οι αποκλήσεις στην εθνική νομοθεσία καταλήγουν σε ανισόρροπη εξέλιξη στις ανανεώσιμες, το οποίο σημαίνει διαφοροποιημένο κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και διαφορετικά επίπεδα εξάρτησης ενεργειακής. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι οι μηχανισμοί στήριξης στα ανανεώσιμα έχουν έναν συγκεκριμένο και απτό αντίκτυπο σε όλες αυτές τις τεχνολογίες ή στην ενέργεια που έχουν και τη δική τους εξέλιξη μερικές φορές τόσο ταχεία που πρέπει να ξαναεξετάσει κανείς ακόμα και την αναγκαιότητα ενός χρηματοδοτικού μέσου στήριξης των τεχνολογιών των ανανεωσίμων. Αυτά τα λέω για να πούμε ότι στηρίζοντας την εισηγήτρια στη βασική της θεωρία χρειαζόμαστε μια πιο φιλόδοξη στόχευση σε ό,τι αφορά στο μέλλον. Απουσία μιας περιφερειοποίησης των μηχανισμών αυτών στήριξης, η πορεία προς την ενσωμάτωση των ε, αναδειωμένων αγορών κινδυνεύει να μείνει ε, εχμάλωτη των ε, περιφερειοποιημένων αν θέλετε συμφερόντων. Χρειαζόμαστε τεχνολογίες ανανεωσίμων που να μην ηλιγήσουν υπό το βάρος του ρυθμιστικού πλαισίου και κυρίως ξένων ανταγωνιστών πιο δυνατών. Μιλάω για τους υδάτινους πόρους και την καλύτερη χρησιμοποίησή τους και ένα καλύτερο σετ κανόνων που χρειαζόμαστε για τα υδροηλεκτρικά που εμεί δεν έχουμε διερευνήσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα επαρκώ. Εκεί χρειάζεται μια πλήρης ένταξη και ενσωμάτωση στις υπόλοιπε ανανεώσιμε πηγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρέδρικ Μπόρλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο ζητήματα με απασχολούν κάπως ως Σουηδό που τα πάμε καλά στις ανανεώσιμες και ενδιαφέρομαι εδώ ιδίως για τη βιομάζα και εννοώ τα κριτήρια της διάρκειας, της βιωσιμότητας. Μπορεί να έχουμε τον ε, τομέα αυτόν υγιή, μπορεί και να τον στραγγαλίσουμε. Υπάρχει παραγωγή βιομάζας και για ηλεκτρικό, για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και για τη θέρμανση αν συνεχίσουμε να ψηφίζουμε σχετική νομοθεσία, μπορεί εν τέλει να ανακόψουμε την πρόοδο αυτή. Δεύτερο, ε, το, η αρχή του cascading, της ε, διαδοχικής ε, δηλαδή διαχείρισης με εταιρείε επί εταιριών. Κάποια εργοστάσια, ιδίως στο Νότο, χάρτου καταναλώνουν 3, ε, ε, παράγουν 3 τεραβάτ ε, ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύουν σε άλλους παραγωγούς. Αν μπορέσουμε να νομιμοποιήσουμε αυτή την αρχή cascading, θα μπορέσουν να διατηρήσουν την παραγωγή που έχουν. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, για παράδειγμα τη Φιλανδία, όπου προχωρούν χρησιμοποιώντας το, τα προϊόντα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για θέρμανση, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, χαρτιού, ακόμη και ε, υφασμάτων για ε, ε, ρουχισμό. Πριν λοιπόν αναλάβουμε οποιαδήποτε ρύθμιση για βιωσιμότητα ε, πηγών ενέργειας όπως το αέριο και ο άνθρακας, να κοιτάξουμε πρώτα τι γίνεται με τη βιομάζα. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Η κυρία Κούμπουλα Νάτρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα σχόλιο για τον Σουηδό συνάδελφο. Το 38% στο παρελθόν είχαμε εμεί, 40% τώρα. ένας λόγος είναι ότι χρησιμοποιούμε τη βιομάζα μας Στόχο νομίζω είναι να έχουμε βιώσιμη βιομάζα και εφόσον υπάρχει αυτή, τότε οι ε, φορείς της αγοράς θα αποφασίσουν πού και πώς θα χρησιμοποιηθεί. Αναμένουμε λοιπόν πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό των κριτηρίων βιωσιμότητας και για την προαγωγή μιας συνεκτικής νομοθεσίας στην Ευρώπη που να ανοίγει πολλές ευκαιρίες και για την ασφάλεια ενέργειας και για το φυσικό αέριο για τη θέρμανση των σπιτιών και ούτω καθεξής. Εξήτασα το κείμενο. Ευχαριστώ την εισηγητρία γιατί είναι ξεκάθαρο, ευανάγνωστο και ευνόητο. Περιλαμβάνει σωστούς στόχους. Με κάποιες ίσως διαφορετικές διατυπώσεις νομίζω ότι περιλαμβάνει και στην παράγραφο 28 που αναφερόταν στη στρατηγική για τα βιολογικά καύσιμα. Έχουμε συμφωνίες, έχουμε το πλαίσιο μέχρι το 2020. Αλλά μετά μιλούν πολύ για την ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική τεχνολογία, αλλά αλλά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μονάχα κατά 26% ανανεώσιμο. Όταν θα έχουμε τις, τους κινητήρες αυτούς που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ε, ορυκτά καύσιμα, γιατί να μην τα βάλουμε και αυτά εκεί. Λοιπόν, τι κάνουμε, παρετούμεθα από αυτό ή εξακολουθούμε να πιέζουμε ώστε να αφαιρεθεί το στοιχείο των εκπομπών διοξιδίων του άνθρακος από τον τομέα των μεταφόρων. Μία σύντομη ερώτηση όμως, Πρόεδρε. Γιατί να μην είναι ε, το ίδιο ε, αποδοτικές και καταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Δηλαδή, γιατί μόνο μικρής κλίμακας. Αν δηλαδή και σε μεγάλη κλίμακα είναι ανανεώσιμες και αποδοτικές οι ενέργειες αυτές, γιατί να είμαστε αντίθετες. Καμιά φορά η οικονομία κλίμακος είναι καλά. Βέβαια, αν είναι και στην Ήπεθρο, ας πούμε, ένα αγρόκτημα κτλ. Η μικρή κλίμακα επίσης είναι καλή. Αλλά να γίνει το ίδιο και για τις, για κέντρα. Ευχαριστώ. Παουλ Ρούμπικ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι στα όσα είπε ο κύριος Ζανονάτο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς θα διαμορφώσουμε αποτελεσματικότερα και την κατανάλωση ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας χρειάζεται και αποθηκευτική ικανότητα, που είναι μία δυνατότητα, μία εναλλακτική επιλογή. Η άλλη εναλλακτική επιλογή είναι η διασύνδεση των ευφυών συστημάτων. μεταξύ Βορρά, Νότου, Ανατολής Δύσης διότι μπορεί να μην υπάρχει ε, μια συγκεκριμένη στιγμή αέρας, δηλαδή άνεμος, στο βορρά θα υπάρχει όμως στο νότο. Κάπου θα υπάρχει, κάπου θα λάβει ο ήλιος. Να συνδεθούν λοιπόν τα συστήματα. Ούτε θα συμβαίνει ώστε παντού ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ευρώπη να υπάρχει και άνεμος και να λάμπει ο ήλιος. Επίσης, οι δυνατότητες αποθήκευσης της ενέργειας είναι σημαντική και χαίρομαι διότι προβλέπεται ακρόαση από την δυνατότητα αποθήκευσης της ε, υδραυλικής ενέργειας μέχρι και των άλλων ενεργειών. Και να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε και μία αγορά για τις αποθηκευτικές ικανότητες της ενέργειας. Χθες βρεθήκαμε στην European Space Agency στις κάτω χώρες. Και κατά την μετάβασή μας εκεί σκέφτηκα το εξής. Γιατί δεν μπορούμε να μειώσουμε τα διοξίδια του άνθρακος και στις μεταφορές, διότι περάσαμε από πραγματικό ερυθρό κύμα, αντί πράσινο κύμα που ανάβουν οι πράσινοι σηματοδότες, είχαμε μπροστά μας διαρκώς ερυθρού κόκκινους σηματοδότες, κόκκινα φανάρια. Πρέπει να είναι ρευστή τι η κυκλοφορία. Να προωθήσουμε πραγματικά το πράσινο κύμα στην Ευρώπη, στην κυκλοφορία εννοώ των αυτοκινήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λιμπής. Τέλος. Ο κύριος Κόχλιτσεκ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Μια παρατήρηση σχετικά με το ότι δεν είμαστε μόνο Επιτροπή Βιομηχανίας, αλλά και τεχνολογίας. Και εδώ στην έκθεση δεν μιλούμε για τεχνολογικά θέματα και για τη στήριξη των τεχνολογικών εξελίξεων. Για τα φωτοβολταϊκά η αποδοτικότητα είναι της τάξης του 11%. Πάρα πολύ χαμηλή. Όμως ήδη σήμερα Υπάρχουν νέες τεχνολογικές μέθοδοι για την αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων αυτών και μάλιστα να διπλασιαστεί. Αυτά βέβαια μπορούν να περιληφθούν σε άλλη έκθεση. Ωστόσο, θα ήθελα στο μέλλον να υποστηρίξουμε τις εξελίξεις αυτές. Τώρα, η αποκέντρωση στους ιδιωτικούς επενδυτές δεν είναι βέβαια το ιδεώδες αυτό. Μικρότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές, σωστό. Όμως, οι δαπάνε για τις ανανεώσιμες ενέργειες αυτές να βαρύνουν τι εθνικές κυβερνήσεις. Γιατί αυτά συνεπάγονται φορολόγηση και η φορολόγηση είναι αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Την στήριξη βέβαια για τους στόχους τη συμμερίζομαι. Αλλά αν έχω ένα ηλεκτρικό όχημα το οποίο τροφοδοτώ από ανανεώσιμε ενέργειε, να μην είναι μόνο εν μέρη, αλλά είναι 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μου χρειάζεται απαραίτητα ένα παραδοσιακό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας για να φορτίσω τις μπαταρίες του αυτοκινήτου μου, τις σωρευτές του αυτοκινήτου μου. Εάν μπορώ να έχω ένα σύστημα το οποίο να καλύπτει τι σε ηλεκτρικό ρεύμα ενός νοικοκυριού, αυτό κοστίζει γύρω στις 10.000 ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε αρκετά εργοστάσια υδραυλικής ενέργειας, είναι αλήθεια, υπάρχει και δυσκολία αποθήκευσης της ενέργειας αυτής, οι δε είναι οι που διαθέτουμε είναι περιορισμένης ικανότητας. Άρα έχουμε ακόμα σημαντικές ελλείψεις. Νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να εγκύψουμε σε αυτά στο περιεχόμενο μια έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια, η Διευθύντρια κυρία Μαρή Ιντόνομη. Και πάλι ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του ευρωβουλευτέ που έδειξαν αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Όπω και τι προηγούμενε φορέ, πρέπει να πω ότι είναι πολύ επίκαιρο γιατί όπω ξέρετε εξετάζουμε την αναθεώρηση ε, της οδηγίας ΑΠΕ μέχρι τα τέλη τη χρονιά. Και πολλά από τα θέματα που έχετε συμπεριλάβει στο σχέδιο έκθεσή σα και αναφέρατε και στη σημερινή συζήτηση είναι ζητήματα που μας απασχολούν και εμά. Για να σταθώ σε ορισμένα από τα σχόλια που ακούσαμε. Η εμπιστοσύνη ε, των ε, επενδυτών είναι σημείο κλειδί σε αυτό το κλάδο γιατί είναι ε, απαιτητικέ σε κεφάλαια οι ΑΠΕ και αυτή τη στιγμή δεν έχουν ενταχθεί πλήρως στις τιμές της αγορά. Γι' αυτό και η στήριξη από πλευρά πολιτικής δεν εντάσσεται απαραίτητο στον τομέα των ΑΠΕ, αλλά θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο. Τέτοιου είδους ε, στήριξη θα πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο ε, για τη γεφύρωση του χάσματος του επενδυτικού στις ΑΠΕ, αλλά και για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην αγορά. Αλλά και για την ε, μετάπτωση την ενεργειακή. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για την αναθεώρηση της οδηγίας οι διατάξεις για τις συνοδευτικές προτάσεις, ETS πέρυσι και ανασχεδιασμός τη αγοράς φέτο, όλα αυτά θα συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η οδηγία παρουσιάζει μια ευκαιρία προβολής και επιβεβαίωση του ρόλου του πολίτη και του καταναλωτή στο επίκεντρο του ενεργειακού συστήματο. Και ω προ αυτή την άποψη έχουμε και το πολύ σημαντικό ρόλο των παραγωγών καταναλωτών και τη αποκεντρωμένη παραγωγή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε και να λάβουμε υπόψη στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης. Κέριο ζήτημα, και σας ευχαριστώ που το θίξατε, είναι ότι οι ανανεώσιμε βεβαίω διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως θα πρέπει στη συνέχεια να διαδραματίζουν και πολύ σημαντικό ρόλο και σε ό,τι αφορά τη θέρμανση και ψήξη, 50% της καταναλωση ενέργειας, αλλά και στον τομέα των μεταφορών. Είναι σημαντικό αυτές οι δυνατότητες να προβάλλονται και να στηρίζονται και πολιτικά ως προς την προώθηση των δραστηριοτήτων μας σε αυτό το τομέα και σας ευχαριστώ που τα αναφέρετε ρητός ε, στην έκθεση. Χρηματοδοτικός μηχανισμός για τις ανανεώσιμες. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει χρηματοδοτικό χάσμα γιατί ε, είναι πολύ απαιτητικέ σε κεφάλαια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκή κίνητρα στην αγορά Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους ε, χρηματοδοτικός μηχανισμός για την μείωση του ε, κινδύνου, του ρίσκου. Είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Ε, ε Βεβαίω στηρίζουμε και τις εξελίξεις στην έρευνα και καινοτομία. Υπάρχει και ο αντίστοιχο οδικό χάρτη στον του 2020. Εκεί έχουμε συγκεκριμένα αναφέρει την αποθήκευση ω ε, κύριο στόχο ε, για όλου του τομεί, ε, την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων και την ανταπόκριση με βάση τη ζήτηση. Και αυτό συνδέεται στενά και με τι προηγούμενε συζητήσει για την ενεργική απόδοση. Νομίζω ότι έχουμε δύο στοιχεία προβληματισμού, τα οποία επίσης έχουν αναφερθεί σήμερα το απόγευμα. Έχουμε την, τα κριτήρια βιωσιμότητα στη βιοενέργεια. Είναι κάτι ή μάλλον τα υφιστάμενα ε, κριτήρια θεωρούμε ότι είναι τα καλύτερα στον κόσμο που προβλέπονται από τη σημερινή οδηγία. Βεβαίω και μπορούν να βελτιωθούν και σκοπεύουμε να το κάνουμε. Αλλά με έναν τρόπο που να αντικατοπτρίζει την ε, πολύ λεπτή ισορροπία που έχουμε πετύχει ήδη στο κείμενο και τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την σωστή διαχείριση των βιοκαυσίμων και της βιοενέργειας στις οικονομίες μας. Δεύτερο στοιχείο προγραμματισμού, οι μεταφορές. Μεγάλη πρόκληση το μέσα των μεταφορών πολλέ δυσκολίε. Το έχουμε συζητήσει και εδώ στο Κοινοβούλιο και γενικότερα εδώ στι Βρυξέλλε. Όλο αυτό το θέμα τη βιοενέργεια στι μεταφορέ. Καταλήξαμε συμπεράσματα πέρυσι. Παραμένει όμω η πρόκληση, αλλά και η ευκαιρία να κάνουμε κάτι στο δομέα των μεταφορών με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων. Και αυτό είναι ένα, ένα από τα θέματα που θα μα απασχολήσουν και στην αναθεώρηση τη οδηγία για τι ανανεώσιμε, αλλά και στην ανακοίνωση για ε, την αποδέσμευση από τον άνθρακα στι μεταφορέ που θα δημοσιευτεί το καλοκαίρι από την Κομισιόν. Σα ευχαριστώ και επιβλέπουμε σε οριστικοποίηση των εργασιών μα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παλώμα Λόπεθ Βερβέχο, εισηγητρία, έχει το λόγο. Eh, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις τους. Μία πτυχή που μου φαίνεται σημαντικό να υπογραμμίσουμε. Τα βιοκαύσιμα. Είναι θα είναι η Επιτροπή Ένβη που θα αναπτύξει το στοιχείο αυτό, είναι αρμοδιότητά της. Εδώ μιλούμε για μια γενική ανάλυση, απλώς, και ελπίζω να μπορέσουν οι πολιτικές ομάδες να την στηρίξουν. Είναι η τρίτη φορά που συναντιόμαστε για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Εγώ σημείωσα προσεκτικά όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν σήμερα Και βεβαίω ε, εξετάζουμε και συνεχίζουμε, να εξετάζουμε τις 345 τροπολογίε. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχετε συμβαστικό κείμενο που είμαι βέβαιη ότι θα ενσωματώνει πολλές από τις τροπολογίε αυτές και με αυτό είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε πιο εύκολα <clears throat> να επιτύχουμε μια συμφωνία. Με ευρύτατη πλειοψηφία θέλω να πιστεύω. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Σας ευχαριστώ εκ νέου για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια, λέει ο Πρόεδρος. για τα σχόλιά της και ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά τους. 24 Μαΐου στην Ήτρε και ψήφος στην Ολομέλεια στη δεύτερη Ολομέλεια του Ιουνίου Και με αυτό ολοκληρώσαμε τη διάταξη για σήμερα, το απόγευμα, για τους περισσότερους βέβαια, αλλά όχι και για τους συντονίστες, για τους οποίους, από τους οποίους χρειαζόμαστε ακόμα μία ώρα. Για τους υπόλοιπους θα συναντηθούμε στις 9 το πρωί την επόμενη φορά και έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Πολιτισμού 7 με 9 το βράδυ τη Δευτέρα 9 Μαΐου στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ.